Hello to everybody. Good morning. Καλημέρα σε όλους. Hello. Buongiorno a tutti e a tutte. Καλημέρα σε όλους και όλες και κυρίως σε όλες. Μεγάλη μου χαρά να κηρύξω την έναρξη των εργασιών αυτής της διάσκεψης. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας, τους προσκεκλημένους, τους βουλευτές, τους δημοσιογράφους που βρίσκονται σήμερα εδώ και θα ήθελα λίγα λόγια να εξηγήσω το στόχο αυτής της διάσκεψης σήμερα. Πριν από λίγους μήνες αποφασίσαμε να διοργανώσουμε αυτή τη διάσκεψη με έναν διπλό στόχο. Πρώτον, να κάνουμε έναν απολογισμό των κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή να εξετάσουμε την ευρωπαϊκή παραγωγή οδηγιών, τις οποίες επεξεργάστηκε το Ευρωκοινοβούλιο για θέματα ισότητας φύλου. Και δεύτερο στόχο, να Μικρύνουμε τις αποστάσεις ανάμεσα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τα εθνικά κοινοβούλια και τους πολίτες. Γιατί συμβαίνει που και που τα θεσμικά όργανα να δουλεύουν πολύ, <laughs> να παράγουν πολύ σημαντικές νομοθεσίες, αλλά οι πολίτες να μην έχουν συμμετάσχει επαρκώς, ούτε να έχουν ενημερωθεί επαρκώς. Γι' αυτό και αισθανθήκαμε αυτή την ανάγκη εμπλοκής των συμπολιτών μας ε, να προσπαθήσουμε να έρθουμε πιο κοντά ως θεσμοί στους πολίτες και να τους ενημερώνουμε όσο γίνεται περισσότερο να μπορούν να συμμετέχουν και να γνωρίζουν και τα δικαιώματά τους. Αυτή η διάσκεψη λοιπόν διοργανώθηκε από την ομάδα υψηλού επίπεδου για την ισότητα των φύλων και τη διαφοροποίηση του οποίου είμαι πρόεδρος, η ομάδα επικοινωνίας του Προεδρείου του Ευρωκοινοβουλίου. Αργότερα θα έρθουν δύο αντιπρόεδροι που θα παρέμβουν ε, σε σχέση με την ε, ανακοίνωση για την ισότητα των φύλων και έχουμε και ιδιαίτερη στήριξη από την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και πιο συγκεκριμένα από τον πρόεδρο αυτής, τον κύριο Γκούσταυσον που βλέπετε εδώ στα αριστερά μου. και που είναι ένας εξαιρετικός πρόεδρος. Και δίνει μεγάλη όθηση στην Επιτροπή coloro che si sono resi disponibili Έχετε επίσης στη διάθεσή σας ε, τεκμηρίωση πολύ. Παρακαλώ να δείτε όλα αυτά τα έγγραφα. Ο Γενικός, ε, η Γενική Διευθύντρια Επικοινωνίας η Γιωχάννα Λαούς, ε, ε, ο κύριος Ρικάρντο Ριπέρα, που η Γενική Διεύθυνση της, του, της Προεδρίας με την ειδική της Διεύθυνση για τις σχέσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους ιδιαιτέρως τον αναπληρωτή τη Γενική Γραμματέα, αναπληρώτρια μάλλον Γενική Γραμματέα, την κυρία Φραντσέσκα Αράτη, την Γενική Διεύθυνση Διερμηνίας και Μετάφρασης και μεταξύ άλλων να θυμίσω πως αυτό, αυτή εδώ η διάσκεψη μπορεί να ε, μάλλον αναμεταδίδεται στο ίντερνετ οι ευρωβουλευτές που είναι παρόντες μπορούν ως συνήθως να ζητήσουν το λόγο και οι εθνικοί βουλευτές μπορούν να αναζητήσουν το λόγο δείχνοντάς μας την κάρτα τους με το όνομά τους. Όχι, πρέπει να το φέρουν εδώ. Έχετε ένα χαρτόνι εκεί στην, στα έδρανά σα και αν θέλετε να πάρετε το λόγο θα πρέπει να το παραδώσετε στους κλητήρες που θα το φέρουν εδώ στα έδρανα της Προεδρίας. Να κλείσω λοιπόν αυτή την ε, αναρκτήρια ομιλία διαβάζοντας μια επιστολή που είχε την καλή θέληση ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου μας, Μάρτιν Σούλτσα, να μας διαβιβάσει. Αξιότιμοι κύριοι πρόεδροι, κυρίες ε, ε, βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Σα ζητώ συγγνώμη για την αποσία μου από αυτή τη σημαντική διάσκεψη. Όμω τα καθήκοντά μου ω πρόεδρο του Κοινοβουλίου με οδήγησαν σε, μια, σε κάποιο άλλο κράτο μέλο σε επίσημη επίσκεψη. Θα ήθελα ωστόσο να σα απευθύνω δύο λόγια και να σα καλωσορίσω. Καταρχήν, θα ήθελα προσωπικά να ευχαριστήσω την Επιτροπή ε, για τα δικαιώματα της γυναίκας και την ομάδα υψηλού επίπεδου για την ισότητα και την διαφορετικότητα για αυτή την πρωτοβουλία. Επίσης θα ήθελα να εκφράσω την προσωπική μου γνώμη για το θέμα της ισότητας των φύλων, τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και σε διοικητικό επίπεδο. Η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει την προώθηση της ισότητας ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες ως ρητό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι περήφανος που μπορώ να πω ότι το Ευρωκοινοβούλιο έχει παίξει το ρόλο του και έχει συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου. Η σχέση των γυναικών με την πολιτική, την ισότητα των φίλων ε, φέτος ε, ε, και η σχετική έκθεση που έγινε φέτος οδήγησαν στην πρόθεση αυτών των πολιτικών. Όμως θα πρέπει τώρα να μπουν όλα αυτά σε εφαρμογή μετά από την έγκριση αυτής της έκθεσης στην Ολομέλεια. Η ισορροπία των φύλων θα πρέπει να είναι προνόμιο μόνο των δημοσίων οργανισμών. Ως πολιτική είναι καθήκον μας να προωθήσουμε την ισότητα των φύλων και στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι ένας στόχος ε, για τον οποίο ε, εκμεταλλεύουμε την ευκαιρία και λέω ότι το Ευρωκοινοβούλιο περιμένει με μεγάλη ανυπομονησία να λάβει εντός ολίγου τη σημαντική πρόταση της Κομισιόν για τη βελτίωση της ισών στα συμβούλια των εταιριών που είναι εγγεγραμμένες στο χρηματιστήριο. Αυτό θα συμβάλλει στο να μειωθούν οι, οι, επίμονες ανισορροπίες σε φύλων στα συμβούλια επιχείρηση των εταιριών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιστρέφοντα στο ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο, θεωρώ πω είναι καθήκον μα να δώσουμε το παράδειγμα όσον αφορά την πρόθεση δε των γυναικών στην πολιτική και στο δικό μα θεσμικό όργανο. Τα πολιτικά κόμματα έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στο εθνικό. Επί τη βάση του κανονισμού του Ευρωκοινοβουλίου, στην ε, σημερινή του εκδοχή, Ευρωβουλευτές ε, εκλέγονται μετά από διορισμό των πολιτικών ομάδων. Ανάλογα με τα διάφορα καθήκοντα των αντιπροέδρων και των κοσμητόρων, οι διορισμοί μπορούν να γίνονται μόνο από ε, μια πολιτική ομάδα. Από τη διοικητική πλευρά έχουν ολοκληρωθεί σημαντικά βήματα, αλλά έχουμε ακόμα κάποιο δρόμο να κάνουμε για να υπάρξει ισορροπία φύλων μέσα στο πλαίσιο της Γραμματείας του Ευρωκοινοβουλίου η Προεδρία του Ευρωκοινοβουλίου ως αρμόδιο όργανο που είναι υπεύθυνο για τα θέματα του προσωπικού. Ρητός στήριξε αυτή τη διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη και έχει εγκρίνει το 2006 μια δήλωση για τις αρχές που σχετίζονται με την προώθηση της ισότητας και την διαφορετικότητα μέσα στην γραμματεία. Και το 2009 ένα σχέδιο δράσης για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της διαφορετικότητας έχει εγκριθεί. Κάποιοι στόχοι ισότητας οι οποίοι έχουν οριστεί από το Προεδρείο έχουν επιτευχθεί όσον αφορά ορισμένα τμήματα του προσωπικού. Το 1 τρίτο των γενικών μας διευθυντών και γύρω στο 1 τρίτο των διευθυντών αποτελείται από γυναίκες. Ε, ωστόσο, είμαστε ακόμα πίσω όσον αφορά την γυναική εκπροσώπηση στην ε, ενδιάμεση, στα ενδιάμεσα επίπεδα της διοίκησης. Πάντως το Προεδρείο θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει αυτή την έλλειψη για το υπόλοιπο της θητείας του. Θα ελπίζω τέλος ότι αυτή η κοινή διάσκεψη θα συμβάλλει στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και θα οδηγήσει σε καρποφόρες συζητήσεις. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, Μάρτιν Σούλτ. Ε, Μετά από την επιστολή του και Πρόεδρου Σούλτ θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο Γκούσταυσον. Θυμίζω ότι είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Ευρωκοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Αντζελίδη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Αντζελίλη και τις άλλες αντιπροέδρους της Επιτροπής ε, για τα Δικαιώματα των Γυναικών, τις άλλες αντιπροέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι παρόντα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρήκατε το χρόνο να είσαστε παρόντες και παρούσες σε αυτή τη συνεδρία. Είναι μια μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι δίπλα στην κυρία Αντζελίλη και να συμπροεδρεύω αυτήν την συνδιάσκεψη. Θέλω σας ευχαριστήσω λοιπόν και για την ε, πρωτοβουλία που αναλάβατε κυρία Αντζελίλη για τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε ένα τέτοιο, μια τέτοια κοινή ε, διοργάνωση μεταξύ της ομάδος για την ε, ισότητα ευκαιριών μαζί με την Επιτροπή για τα δικαιώματα των γυναικών και την ίση εκπροσώπηση των φίλων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η συνδιάσκεψή μας είναι μια θαυμάσια ευκαιρία για όλους μας να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε απόψεις μεταξύ μας, να εξηγήσουμε τις εμπειρίες που έχουμε συλλέξει και να μπορέσουμε να έχουμε μεταλαμπάδευση βελτίστων πρακτικών. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό διότι διατρέχουμε μια περίοδο κρίσης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι φανερό ότι η κρίση και οι συνέπειές της έχουν πλήξει ιδιαίτερα τις γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερα στο χώρο της εργασίας όπου οι γυναίκες έχουν χάσει θέσεις εργασίας, έχουν υποστεί τις συνέπειες των περικοπών σε ό,τι αφορά το κοινωνικό κράτος και αναμένουν όλοι εν ώψη αυτών των περικοπών οι γυναίκες να είναι αυτές οι οποίες θα καλύψουν το κένο και το χάσμα το οποίο δημιουργείται. Επομένως εμπλέκονται ιδιαίτερα οι γυναίκες στην Ευρώπη ε, σε μια κατάσταση κρίσης όπως η σημερινή γιατί πάρα πολλέ φορέ αντιμετωπίζεται η κρίση σαν ένα τεχνικό και οικονομικό θέμα, αλλά σε ανθρώπινο επίπεδο είναι κάτι το οποίο εμπλέκει ιδιαίτερα τις γυναίκες. Έχουμε ένα ευρύ πρόγραμμα σήμερα το οποίο θα μας απασχολήσει. Έχετε και στα αναχείρα σα το πρόγραμμα αυτό. Αλλά θέλω να τονίσω ότι έχουμε σήμερα να αντιμετωπίσουμε μια ιδιαίτερα σημαντική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την έκθεση της κυρίας Πιετικάινεν για την ενίσχυση της θέσεως των γυναικών στον πολιτικό στίβο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και υπάρχει μια ευρεία συνένεση μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορέσουμε να εξεύρουμε τα μέτρα μέσω των οποίων θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε την παρουσία των γυναικών στον πολιτικό χώρο. Η κυρία Πιετικάινεν θα είναι παρούσα το απόγευμα και θα μας παρουσιάσει λεπτομεριακά την έκθεση αυτή. Προηγουμένως όμως θέλω να σας αναφέρω το εξής, ότι για διαφόρους λόγους είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχουν γυναίκες σε υψηλά επίπεδα λήψης αποφάσεων. Γι' αυτό μπορεί κανείς να εκφράσει την έλλειψη ικανοποίησής του για γεγονότα όπως το γεγονός ότι πρόσφατα για μια θέση στο Προεδρείο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δεν υπήρξε καμία γυναίκα η οποία είχε προταθεί για τέτοια θέση. Και αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι δεν υπάρχουν γυναίκες οι οποίες είναι ικανές να αναλάβουν αυτό το αξίωμα. Αυτό είναι προφανώς κάτι το οποίο ισχύει. Αλλά δεν υπήρξε καμία υποψήφιος η οποία παρουσιάστηκε για αυτή τη θέση. Η Επιτροπή μου ενδιαφέρεται ιδιαίτερα στο να ενισχύσει τη σχέση και τη σύνδεση με τα Εθνικά Κοινοβούλια και να συζητήσει για το σύνολο αυτών των θεμάτων. Εγώ χαίρομαι λοιπόν για την ευκαιρία να έχουμε και από το Γερμανικό Κοινοβούλιο μια ομάδα επισκεπτών και επίσης και επισκέπτες που έχουν κληθεί από την κυρία Λάουρετσεκ. Νομίζω ότι θα είναι και για αυτούς επωφελείς οι συζητήσεις οι οποίες θα λάβουν χώρα σήμερα. Για μας, τονίζω και πάλι, είναι πάρα πολύ σημαντική η σημασία των στενών επαφών με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Εν κατακλείδη, θα ήθελα να σας πω το εξή, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει το Ινστιτούτο για την ε, ισότητα των φίλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μπορεί να σας παράσχει υλικό, τεκμηριωτικό και να σας δώσει πληροφορίες. Εάν θέλετε θα μπορούσατε να έρθετε σε επαφή με τους εκπροσώπους αυτού του Ινστιτούτου που έχουν συλλέξει στοιχεία, έχουν κάνει έρευνες, έχουν αναπτύξει ερευνητικά προγράμματα. Έχουμε τις ε, επιστημονικές λοιπόν αυτές εμπειρογνωμοσύνες αυτού του Ινστιτούτου που είναι ιδιαίτερα χρήσιμες. Σας ευχαριστώ και πάλι λοιπόν για την παρουσία σας. Ελπίζω ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ καρποφόρα ημερίδα συζήτησης για τα θέματα ισότητας των φίλων Και σας ευχαριστώ που ήρθατε. Grazie, ehm, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ τώρα θα ήθελα να σας παρουσιάσω ένα σύντομο πλαίσιο για τις ε, εργασιακές προοπτικές εντός του προσωπικού του Ευρωκοινοβουλίου. Αυτό είναι σημαντικό γιατί όπως θύμιζε ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου στην επιστολή του, καταρχήν τα θεσμικά όργανα είναι αυτά που πρέπει να δώσουν το καλό παράδειγμα. Είναι πραγματικά άσχημο για ένα κοινοβούλιο και κυρίως για το Ευρωκοινοβούλιο να δίνει κατευθύντριες γραμμές πολιτικής φύσης, ρυθμιστικής φύσης και έπειτα να μην τις εφαρμόζει επί του ίδιου του, του προσωπικού. Άρα λοιπόν είναι ενδιαφέρον να δούμε τη δουλειά που έχει γίνει από την Γενική Διεύθυνση Προσωπικού που μας δίνει ένα πλαίσιο της κατάστασης εντός του ευρώ. Και θα σας δώσω κάποια στοιχεία να καταλάβετε καλύτερα που βρισκόμαστε. Το σύνολο του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το 41,5% των υπαλλήλων είναι άνδρες, ενώ οι γυναίκες είναι το 58,5%. Άρα, εντός του προσωπικού του Ευρωκοινοβουλίου, όντως οι γυναίκες είναι περισσότερες, είναι η πλειοψηφία. Όμως, είναι ενδιαφέρον να αναλύσουμε αυτές τις, ε, αυτά τα στοιχεία από την άποψη της σταδιοδρομίας που ακολουθούν. Η διοίκηση διαιρείται σε δύο τομείς σταδιοδρομίας. Δηλαδή, έχουμε τη σταδιοδρομία ΑΔ, που είναι το διοικητικό προσωπικό, είναι τα πιο, οι πιο υψηλόβαθμοι, 51,3% είναι, είναι γυναίκες και 48,8% ε, με είναι άνδρες. Πάλι έχουν την πλειοψηφία οι γυναίκες. Αλλά μετά θα δούμε καλύτερα σε τι αντιστοιχεί αυτό το νούμερο. Πολύ ενδιαφέρον είναι αντίθετα το νούμερο που αφορά τους βοηθούς και το προσωπικό, το διοικητικό που ονομάζεται AST. Εδώ το 58,5% είναι γυναίκες, ενώ το 41,5% είναι άνδρες. Αυτό τι σημαίνει ότι Είναι αλήθεια ότι οι γυναίκες στο Ευρωκοινοβούλιο και στο προσωπικό του Ευρωκοινοβουλίου είναι η πλειοψηφία, αλλά κυρίως είναι η πλειοψηφία στις μεσαίες και στους μεσαίους και χαμηλούς βαθμούς. Στους χαμηλότερους βαθμούς δε έχουν πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Ενώ στις ψηλότερες θέσεις έχουμε πλειοψηφία γυναικών, αλλά μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο, δηλαδή μέχρι τον βαθμό που ονομάζεται AD8. Δηλαδή είναι ο βαθμός που στην ουσία είναι κάτω από τους τμηματάρχες και όσους θέλουν να ακολουθήσουν ε, πιο στα ε, σταδιοδρομία στο Ευρωκοινοβούλιο. Αν δούμε λοιπόν πιο συγκεκριμένα τα στοιχεία, θα δούμε ότι ανάμεσα στους τμηματάρχες το 74,5% είναι άνδρες και μόνο το 25,5% γυναίκες. Εάν δεν ανέβουμε περισσότερο και φτάσουμε στους διευθυντές, υπάρχει μια μικρή βελτίωση, αλλά πάντοτε έχουμε 67,4% άνδρες και ενώ 32,6% γυναίκες. Αν ανεβούμε δε στο βαθμό των γενικών διευθύντων έχουμε 7 άνδρες προς 4 γυναίκες, δηλαδή 63,6% άνδρες έναντι 36,4% γυναίκες. Και θα ήθελα να διευκρινίσω ότι τα στοιχεία αυτά είναι στοιχεία τα οποία δείχνουν σαφώς βελτίωση σε σχέση με τα τελευταία πέντε χρόνια. Γιατί όπως αναφερόταν και στην επιστολή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, από το 2006 υπήρξε μια πολύ σαφής και ξεκάθαρη δέσμευση από την Προεδρία του Ευρωκοινοβουλίου όσον αφορά την αξιοποίηση των γυναικών. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια είδαμε για πρώτη φορά ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας να είναι γυναίκα, η Φραντσέσκα Ράτη. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της, του Ευρωκοινοβουλίου που μία γυναίκα φτάνει σε ένα τόσο ψηλό βαθμό. Κάτι έχει γίνει λοιπόν. Όμως τα στοιχεία τα οποία μόλις σας έδειξα, σας ανέφερα, είναι ότι ναι μεν οι γυναίκες είναι η πλειοψηφία του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, αλλά περισσότερο είναι πλειοψηφία στις χαμηλόβαθμες θέσεις, ενώ όσο αυξάνονται οι, οι βαθμοί, όσο προχωράει δηλαδή η σταδιοδρομία, βλέπουμε να επικρατούν οι άνδρες. Ρωτήσαμε λοιπόν για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η δυσκολία πρόσβασης στις πιο υψηλόβαθμες θέσεις. Γι' αυτό γιατί πολλές γυναίκες δεν ζητούν καν, δεν υποβάλλουν καν το αίτημα για να φτάσουν σε πιο υψηλόβαθμες θέσεις. Δηλαδή υπάρχει κατά κάποιο τρόπο μια ένα πάγωμα. Δεν θέλουν να πάνε σε ψηλότερες θέσει. Και αυτό γιατί, γιατί και στο εσωτερικό του, της διοίκησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βασικός λόγος για τον οποίο οι γυναίκες <coughs> δεν διεκδικούν περαιτέρω άνοδο στα διδρομία τους είναι η δυσκολία συνδυασμού, συμφιλίωσης του προσωπικής ζωής, της οικογενειακής ζωής με την επαγγελματική. Οι πιο υψηλόβαθμες θέσεις ε, χρειάζονται περισσότερη ε, ε, βοήθεια. Υπάρχει μέσα στο κοινοβούλιο δομή για την φροντίδα των παιδιών, υπάρχει συμπαράσταση και στήριξη στους γονείς. Υπάρχουν διάφορες εγγύησει για την στήριξη της, γυναίκας, της εργαζόμενης γυναίκας, όμως υπάρχει ένα μια οροφή, μια οροφή κρυστάλλινη όπως αποκαλείται, που εμποδίζει τις γυναίκες να προχωρήσουν ακόμα και όταν θα μπορούσαν να το κάνουν από πρακτική άποψης. Γιατί, γιατί πέρα από ένα κάποιο συγκεκριμένο όριο η γυναίκα δεν έχει τη διάθεση να εγκαταλείψει αυτές τις ε, θέσεις το 55% των γυναικών που ερωτήθηκαν απάντησαν ότι δεν διεκδικούμε ψηλότερε θέσει γιατί είναι δύσκολο να συνδυάσουμε την εργασιακή ζωή με την οικογενειακή. Βεβαίω, οι καταστάσει διαφέρουν. Μπορεί να υπάρχουν παιδιά, μπορεί να υπάρχουν ε, ηλικιωμένοι, μπορεί να υπάρχουν ε, ανάπηροι. Μπορεί να υπάρχουν μονογονεϊκές οικογένειες, όπως λέγονται, που η γυναίκα είναι ο αρχηγός της οικογένειας και η μόνη η οποία ασχολείται ίσως με τα παιδιά που έχει για τα οποία είναι υπεύθυνη. Είναι ενδιαφέρον λοιπόν να δει κανείς ότι ακόμα και σε ένα τέτοιο εργασιακό περιβάλλον όπως αυτό το Ευρωκοινοβουλίου ο πρώτος λόγος, ο πρώτος φραγμός σε σχέση με την πρόοδο στη σταδιοδρομία είναι η συμφιλίωση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή. Ρωτήσαμε μετά τα κράτη-μέλη, τα εθνικά κοινοβούλια, αν είχαν στον εσωτερικό τους κανονισμό συγκεκριμένες στρατηγικές για το προσωπικό των κοινοβουλίων. Και τα εθνικά κοινοβούλια μας απάντησαν. Μόνο τέσσερες, τέσσερις βουλές έχουν συγκεκριμένα προγράμματα για το γυναικείο τους προσωπικό. Γερμανία, Ουγγαρία, Φιλανδία και Γερμανία. Είναι οι μόνες χώρες και Ολλανδία, με συγχωρείτε. Είναι οι μόνες χώρες όπου υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα για τις γυναίκες εργαζόμενες. αυτά για τα εθνικά κοινοβούλια. Είναι ανησυχητικό αυτό το στοιχείο. <laughs> Α, δείτε ότι είμαστε 27 κράτη-μέλη και μόνο τα τέσσερα σκεφτήκαν ειδικά προγράμματα για τις γυναίκες στα κοινοβούλια τους. Και γιατί είναι αρνητικό αυτό, διότι αν οι θεσμοί, δηλαδή σε αυτή την περίπτωση τα κοινοβούλια, αυτοί δηλαδή οι οποίοι συντάζουν τις νομοθεσίες, εκδίδουν κανόνες, δίνουν οδηγίες και δεν τηρούν αυτές τις ίδιες τις οδηγίες σε μια φάση, ειδικά σε μια φάση οικονομικής κρίσης, ο ιδιωτικός κόσμος, οι ιδιωτικές εταιρείες, τι θα κάνουν, θα προσπαθήσουν να ξεφύγουν από τις υποκρεώσεις αυτές. από τα προγράμματα που ευνοούν δηλαδή την πρόοδο των γυναικών στη σταδιοδρομία. Επιστρέφω λοιπόν στην επιστολή του Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου που έλεγε ότι τα θεσμικά όργανα έχουν την υποχρέωση να δίνουν το καλό παράδειγμα γιατί διαφορετικά είναι πολύ πιο δύσκολο να επιβληθούν οι κανόνες όταν ε, δεν μπορεί κανείς να αυτορυθμιστεί με τρόπο υποδειγματικό, αποτελεσματικό, με έναν τρόπο δηλαδή που να μας επιτρέπει όλες να εξηγήσουμε γιατί οι γυναίκες πρέπει να έχουν την ευκαιρία να σταδιοδρομήσουν και να είναι επίσης ώρες με τους άνδρες, αν το επιθυμούν. Επιπλέον σε αυτά θα ήθελα να προσθέσω κάποια στοιχεία τα οποία ήδη προανέφερα χτες σε ένα σεμινάριο με τους ε, δημοσιογράφους. Ήθελα να δώσω κάποια στοιχεία για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, να περάσουμε δηλαδή από, από το προσωπικό στους ευρωβουλευτές, τους ερετούς εκπροσώπους των λαών εντός της Ευρωπαϊκής, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί να το κάνω αυτό, γιατί τα στοιχεία πιο γλαφυρά μας δίνουν ε, την εικόνα της πραγματικότητας. Ας ξεκινήσουμε από την Ευρωπαϊκή Εκτελεστική Επιτροπή. 12 πρόεδροι είχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τώρα και ούτε ένας από αυτούς δεν ήταν γυναίκα. Ο πρόεδρος Γκούσταυσον μας θύμισε μάλιστα εχθές ότι στο εσωτερικό της ε, ΕΚΤ, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δεν υπάρχει ούτε μία γυναίκα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μάλιστα εχθές, ε, ε, καλώντας τους συναδέλφους της αυτή εδώ τη διάσκεψη, μια συνάδελφος αστευόμενη μου στείλε ένα mail με τη φωτογραφία των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που μιλά πολύ, πιο, πολύ περισσότερο από, από τα λόγια. Γιατί είναι μόνο άνδρες αυτή τη φωτογραφία. Μια φωτογραφία λέει πολύ περισσότερο από τα λόγια. Ας πάμε τώρα να δούμε το Ευρωκοινοβούλιο. 29 προέδρους έχει αλλάξει το Ευρωκοινοβούλιο, ένα σωρό δηλαδή. Δύο μόνο γυναίκες υπήρξαν πρόεδροι του Ευρωκοινοβουλίου. Η Σιμών Βέιλ και η Νικόλ Φοντέν. 2 στις 29. Να μην αναφέρω σε ποσοστό πόσο μας κάνει αυτό. 2 στις 29. Τώρα, επίσης για το Ευρωκοινοβούλιο να πω ότι Από το 1979, δηλαδή από την πρώτη φορά που εξελέγησαν ευρωβουλευτές στο Ευρωκοινοβούλιο, οι γυναίκες τότε ήταν μόλις το 17% των ε, ευρωβουλευτών. Το 1979, 30 χρόνια μετά, με τούτη εδώ τη θητεία έχουμε κλείσει τα 30 χρόνια, δηλαδή το 2009, οι γυναίκες αντιπροσωπεύονται ε, κατά 34%. Μας πήρε 30 χρόνια δηλαδή για να διπλασιάσουμε την παρουσία των γυναικών μέσα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Και μάλιστα θα πρέπει να είμαστε και πολύ ικανοποιημένες. Ε, ικανοποιημένοι, διότι εάν δούμε τι γίνεται στα κράτη-μέλη, στα 27 κράτη-μέλη, οι γυναίκες στο εσωτερικό των Εθνικών Κοινοβουλίων είναι κατά μέσο όρο μόλις 25% των ερετών εκπροσώπων, ακόμη πιο χαμηλό ποσοστό δηλαδή. Και αν δούμε τις γυναίκες που έχουν κάποιο κυβερνητικό έργο, είναι υπουργοί δηλαδή στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, αυτό το νούμερο φτάνει στο 23% μόλις. Αυτά τα στοιχεία όλα λοιπόν θα πρέπει να μας κάνουν να σκεφτούμε, να προβληματιστούμε. Είναι πιο δύσκολο να μιλήσουμε στην κοινωνία των πολιτών, στις εταιρείες και να επιβάλλουμε όρια και στόχους όταν τα ίδια τα θεσμικά όργανα δυστυχώς είμαστε πολύ πίσω όσον αφορά την επίτευξη αυτών των στόχων. Ο ίδιος ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου μας έλεγε σε ένα κομμάτι του κειμένου που ίσως να μην ήταν και απόλυτα ξεκάθαρο, μιλώντας για το ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο, έλεγε ότι ο διορισμός των προέδρων των επιτροπών ή των αντιπροέδρων του Ευρωκοινοβουλίου εξαρτάται από τις πολιτικές ομάδες. Δηλαδή, οι ίδιες οι πολιτικές ομάδες είναι αυτές που ορίζουν τους υποψηφίους τους και έπειτα οι επιτροπές του Κοινοβούλιου ψηφίζουν για τους διαφόρους ε, ε, προέδρους ή αντιπροέδρους του Ευρωκοινοβουλίου. Όμως, οι πολιτικές ομάδες σε τούτη τη θητεία έδωσαν ένα πολύ ε, δυνατό χτύπημα στην ισότητα των φύλων. Να σας πω, το 2009 οι γυναίκες αντιπρόεδροι του Ευρωκοινοβουλίου ήταν έξι. Όπως γνωρίζετε μετά από δυόμιση χρόνια γίνεται μια αλλαγή βάρδιας και επαναπροσδιορισμός των αξιωμάτων και οι πολιτικές ομάδες υπέδειξαν όχι πια έξι, αλλά τρεις μόνο. Τρεις μόνο αντιπροέδρους γυναίκες από τους 14. Δείτε σε τι ποσοστά αντιστοιχεί αυτό μόνοι σας. Τώρα, όσον αφορά τους πρόεδρους των επιτροπών, Έχουμε 22 προέδρους ε, επιτροπών και υποεπιτροπών και περάσαμε από τις 10 γυναίκες του 2019 ε, στις 8 του το 2012. Και από εκεί δόθηκε ακόμα ένα χτύπημα. Θα μπορούσα να συνεχίσω να μιλάω και να σας δίνω και άλλα στοιχεία. Αλλά νομίζω πως σας έδωσα αρκετά ήδη για να υπογραμμίσω με αυτόν τον τρόπο πως έχουμε φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο πια που μάλιστα υπογραμμίστηκε ακόμη περισσότερο τις περασμένες εβδομάδες στο πλαίσιο της συζήτησης των ποσοστώσεων. Την πρόταση δηλαδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ποσοστώσεις για τις εταιρείε που είναι γεγραμμένες στο χρηματιστήριο. Όπως ξέρετε, η Επίτροπος Ρέντινγκ πριν από δύο χρόνια περίπου είχε εντοπίσει αυτό το στοιχείο το πολύ ανησυχητικό, ότι δηλαδή συνήθως υπήρχε μία γυναίκα, 13% δηλαδή, ε, σε κάθε συμβούλιο επιχείρησης. τότε είχε κάνει αυτή τη διαπίστωση και ξεκίνησε με βάση με λαβή αυτό το στοιχείο μια ολόκληρη συζήτηση, όχι στοιχειο μια ολοκληρη συζητηση οχι απαραιτητος για εισαγωγή ποσοστώσεων, αλλά γιατί και η ίδια δεν είναι απολύτω υπέρ τη εισήγηση των ποσοστώσεων, αλλά μια συζήτηση για συνεργασία από πλευρά των ευρωπαϊκών εταιριών. Και πίστεψε πολύ σε αυτή την προσέγγιση, την εθελούσια, α πούμε. Όμως, δυστυχώς, τα αποτελέσματα όπως ξέρετε δεν ήταν και πολύ ευχάριστα γιατί μετά από λίγο παραπάνω από ένα έτος οι ευρωπαϊκές εταιρείες οι οποίες προσαρμόστηκαν σε ένα τέτοιο αποδεκτό στάνταρ πρότυπο και που ανταποκρίθηκαν στην έκκληση της, ε, της Επιτρόπου ήταν μόλις 24. Μόνο 24 επιχειρήσεις που είναι στο χρηματιστήριο σε ολόκληρη την Ευρώπη ανταποκρίθηκαν. Φρικτό Τότε λοιπόν η Reading ξεκίνησε αυτή την δημόσια διαβούλευση που ολοκληρώθηκε το περασμένο Μάιο και αποφάσισε να έρθει σε επαφή άμεσα με τις εργαζόμενες, με τις επιχειρηματίες και να προτείνει μια νομοθετική διαδικασία, δηλαδή μια πρόταση οδηγίας για να εισάγει ποσοστώσεις υποχρεωτικά. Ξέρετε ότι αμέσως μετά φτιάχτηκε μια ομάδα κρατών εργασ... Ε, μελών με την δυνατότητα να μπλοκάρουν την, ε, απόφαση και χωρίς να υπάρχει καν κείμενο η Ρέντινγκ είχε απλά ανακοινώσει την πρόθεση για επεξεργασία οδηγία. Δεν υπάρχει ακόμα κανένα έγγραφο ανησυχητικό που να μπορεί να προκαλέσει συγκεκριμένα προβλήματα. Όχι. Μόνο και μόνο η ανακοίνωση ότι μπορεί και να υπάρξει μια τέτοια οδηγία οδήγησε αυτά τα κράτη-μέλη να φτιάξουν μια μειοψηφία ε, που μπορεί όμως να μπλοκάρει. 12 ε, κράτη-μέλη μπορεί να μπλοκάρουν την απόφαση και μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας μπορούν βέβαια τα υπόλοιπα κράτη να δώσουν το καλό παράδειγμα. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να σας πω ότι δεν ήμουν ποτέ ιδιαίτερος υπέρ του συστήματος των ποσοστώσεων, γιατί εγώ είμαι γυναίκα σκεφτόμουν ανέκαθεν ναι, ότι μια γυναίκα, όπως κάθε άνθρωπος, θα πρέπει να προχωρήσει με βάση την αξία της, αξιοκρατικά, με βάση τις δυνατότητές της, το πνεύμα θυσίας, αυτοθυσίας κτλ. Δεν ήθελα δηλαδή να θεωρούμαστε ως ένα απόθεμα ή κάτι διαφορετικό που είναι ε, που εννοείται ότι είναι πιο αδύναμη, λιγότερο έξυπνη και λιγότερο αξιόλογη. Αυτά, αυτά είναι στερεότυπα κατά τη γνώμη μου. Ε, κάλλιστα μπορεί μια γυναίκα να φτάσει σε πολύ ψηλό επίπεδο στη διαδρομία της και να συνδυάσει και την οικογενειακή της ζωή. Ανέκαθεν το πίστευα αυτό. Κατέλαβα όμως μετά από κάποια φάση ότι αυτά τα στερεότυπα υπάρχουν, υπάρχουν ως φραγμοί ως εμπόδια, υπάρχουν βέβαια και αντικειμενικά εμπόδια, η έλλειψη ας πούμε υπηρεσιών που να συνοδεύουν μια γυναίκα να τη στηρίζουν για να συμφιλιώσει την οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή. Ας πούμε μια γυναίκα χωρίς νηπιαγωγείο, χωρίς ε, κάποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες δεν μπορεί να προχωρήσει τη ζωή της με αυτόν τον τρόπο. Αλλά μετά κατάλαβα ότι πέρα από όλα αυτά τα πρακτικά, και ανάμεσα σε όλους αυτούς τους άντρες που αποφασίζουν και μιλήσαμε για πολλούς από αυτούς, μιλήσαμε για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, για τα πολιτικά, ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, για την Κομισιόν, για το Ευρωκοινοβούλιο, που πολιτικά κόμματα που την τελευταία θητεία απέδειξαν ότι όταν είναι για να διαλέξουν τους πιο υψηλά ιστάμενους, διαλέγουν άνδρες. Και ακόμα και αν κάποιος θέλει να πει ότι δεν αξίζουμε και πολλά οι γυναίκες, ε, τα στοιχεία αποδεικνύουν το αντίθετο. Αποδεικνύουν ότι από τον πληθυσμό των Ευρωπαίων πτυχιούχων το 60% είναι γυναίκες. Οι γυναίκες είναι αυτές δηλαδή που είναι πιο δραστήριες όσον αφορά την εκπαίδευση και μάλιστα την ανώτατη εκπαίδευση, την πανεπιστημιακή και μετά από το πανεπιστήμιο είναι αυτές που πρώτες παίρνουν το πτυχίο και έχουν και πιο ψηλούς βαθμούς. Αυτά τα λένε οι στατιστικές, τα λέει η Eurostat, δεν τα βγάζω εγώ από το μυαλό μου. Δεν είναι προσωπική μου άποψη δηλαδή μόνο. Γι' αυτό πιστεύω ότι από αυτό το στοιχείο θα πρέπει να ξεκινήσουμε, από τα δεδομένα, από τα στοιχεία που έχουμε στη διαθεσή μας. Η Reading και σίγουρα σήμερα θα μας το αναφέρει, έχει κάνει και μελέτες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των εταιριών που αξιοποιούν τις γυναίκες και που δίνουν αβαντάζ στις γυναίκες, ότι έχουν δηλαδή βαθμό αριστείας πολύ ψηλότερο και έχουν και καλύτερη στάση απέναντι ας πούμε στη διαφθορά που είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ξεκινούσα λοιπόν από τα θετικά αυτά στοιχεία, θα ξεκινούσα και από τα αρνητικά στοιχεία, δηλαδή από τη λιγοστή παρουσία των γυναικών στα επίπεδα λήψης αποφάσεων, από, την ανεπαρκή, ε, από τις ανεπαρκείς ευκαιρίες συμφιλίωσης επαγγελματικής με οικογενειακή ε, ζωή. Και θα ξεκινούσα λοιπόν από ένα τραπέζι εργασίας, ε, κάτι μέλη, Ευρωκοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γιατί πιστεύω ότι αν καθίσουμε όλοι γύρω από το ίδιο τραπέζι θα μπορέσουμε να φτιάξουμε έναν ενάρετο κύκλο ε, για να μπορέσουμε και να συνεργαστούμε καλύτερα και να ενημερώσουμε καλύτερα τους Ευρωπαίους πολίτες ε, ώστε να συμμετέχουν και να εμπλακούν στις διαδικασίες λήψης απόφασης αλλά και για να τους δώσουμε περισσότερη εμπιστοσύνη. Ένα άλλο δε στοιχείο που θα βρείτε στην τεκμηρίωση που σας έχω δώσει είναι ότι οι γυναίκες όταν ερωτηθούν για το πώς βλέπουν το μέλλον, οι γυναίκες είναι αυτές που είναι οι πιο αρνητικές δυστυχώς. Αρνητικές όχι γιατί είναι ε, σε κατάθλιψη, αλλά γιατί βλέπουν ότι βλέπουν με ανησυχία τις ε, συντάξεις γιατί εξακολουθεί να υπάρχει ας πούμε ανισότητα στις αμοιβέ. Γύρω στο 17% λιγότερο κερδίζουν οι γυναίκες κατά μέσο όρο. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία θα πρέπει κανείς να σκεφτεί. Και έτσι κλείνω. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας παρακαλώ να δείτε, να ρίξετε μια ματιά σε αυτήν την τεκμηρίωση που έχει φτιάξει η γραμματεία μας και που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα γιατί είναι μια πληρέστατη εικόνα της πραγματικότητας και βεβαίως αν υπάρχουν ερωτήσεις, παρατηρήσεις, μαρτυρίες, παρεμβάσεις, με χαρά φυσικά θα τις ακούσουμε. Good morning everyone. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σας. Ε, πρωτού ξεκινήσουμε με τις ανταλλαγές ε, ερωτήσεων και απαντήσεων. Λέγομαι Τίτα Σούλτς, είμαι από την ΚΟΠΕΚ που είναι η εσωτερική υπηρεσία και επιτροπή για την ε, ισότητα ευκαιριών στο διοικητικό επίπεδο. Θα ευχαριστήσω και τους δύο συνδιοργανωτές και την κυρία Αντζελίλη και τον κύριο Γκούσταυσον. και τους ευχαριστώ για την ευκαιρία να κάνω μια σύντομη δήλωση. Τι είναι η ΚΟΠΕΚ. Είμαστε μια μικρή συμβουλευτική υπηρεσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με οκτώ μέλη. Εκπροσωπούμε τέσσερις στην δίκηση και τέσσερις στην Επιτροπή Προσωπικού. Για να σας εξηγήσω σε ποιες συνθήκες εργαζόμαστε, δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένος προϋπολογισμός για μας. Έχουμε συναδέλφους στο Λουξεμβούργο και άλλους Φρυξέλλες. Μόνο με βιντεοδιάσκεψη μπορούμε να συνεννοούμεθα και έχουμε όλοι μας κάποιες άλλες αρμοδιότητες πέραν της ΚΟΠΕΚ. Ο στόχος μας είναι να παροτρύνουμε τη δημιουργία ενός θετικού περιβάλλοντος για την ισότητα των φύλων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το κάνουμε αυτό με γνωμοδοτήσεις που εκδίδουμε σε σχέση με την εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης. Είμαστε παρατηρητές σε διάφορες επιτροπές, όπως αυτή για την ευμάρεια του προσωπικού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή Προαγωγών και την υψηλού επίπεδο ομάδα για την ισότητα και τη διαφορετικότητα συνεργασία. Έχουμε τη δυνατότητα επίσης να ξεκινήσουμε ε, ενέργειες για μεγαλύτερη συνειδητοποίηση και εάν προστρέξει σε μας κάποιο μέλος του προσωπικού μπορούμε να δώσουμε και τα φώτα μας σε ό,τι αφορά διοικητικά θέματα. Το γενικό πλαίσιο για μας είναι το σχέδιο δράσης το οποίο ενέκρινε το Προεδρείο και το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένες πολιτικές δεσμεύσεις. <clears throat> για μας είναι το βασικό πλαίσιο. Υπάρχει μια μπροσούρα την οποία έχουμε στην αίθουσα και η οποία περιλαμβάνει τους στόχους της ΚΟΠΕΚ για το χρονικό διάστημα 2011-2014. Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες προς τις ε, μονάδες για την ισότητα του προσωπικού της Γενικής Διευθύνσης Προσωπικού, που είναι πολύ χρήσιμες στατιστικές που καταρτίζουν και αναφέρθηκαν αυτές οι στατιστικές, τα στατιστικά στοιχεία από τον ε, ε, κύριο Γκούσταυσον και την κυρία Αντζελίλη. Φυσικά, η ΚΟΠΕΚ πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως και όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να είναι πρωτοπόρα και υποδείγματα στον τομέα της ισότητας ευκαιριών. Έχει γίνει κάποια πρόοδος τα τελευταία δέκα χρόνια, αλλά δεν έχουμε ακόμα <clears throat> διατρέξει όλο το δρόμο που χρειάζεται. Αναφέρθηκε το θέμα της απουσίας των γυναικών στα μεσαία στελεχικά επίπεδα και βλέπετε ότι μόνο το 1 τρίτο των μεσαίων στελεχών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι γυναίκε. Η ΚΟΠΕΚ πιστεύει ότι χρειαζόμαστε περισσότερη ευκαμψία στο χώρο εργασία μα πέραν των μέτρων κατάρτιση και δημιουργίας και συνειδητοποίηση για το προσωπικό. Είμαστε ιδιαίτερα λοιπόν ευτυχείς για τη σημερινή ευκαιρία που έχουμε να ανταλλάξουμε απόψει με μέλη από, Ευρωπα, από τα Εθνικά Κοινοβούλια και αναμένουμε τις απόψεις σας και ευχαριστούμε για τις ε, απαντήσεις που μας δώσατε στο ερωτηματολογιό μας και θεωρώ ιδιαίτερα χρήσιμα και ενδιαφέροντα τα μέτρα τα οποία ισχύουν στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο και η Κοπέκ επίσης θα ενδιαφερόταν να ακούσει από εσά αν έχετε ένα τέτοιο αντίστοιχο όργανο, ένα συμβουλευτικό όργανο στο Εθνικό σας Κοινοβούλιο. Εάν όχι ποια ήταν η κεκτημένη εμπειρία από αυτό το όργανο. Επίσης, σε σχέση με τα μέτρα τα οποία εφαρμόζουμε στον τόπο εργασίας για την ισορροπία οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, όλα αυτά τα μέτρα τα χρησιμοποιούν κατά 80% οι γυναίκες, όπως είναι η ημερική ε, απασχόληση, η γονική άδεια ή άλλα. Θα ήθελα να ξέρω αν έχετε και εσείς αντίστοιχες εμπειρίες και αντίστοιχα μέτρα και αν ενθαρρύνετε τους άντρες και αυτοί να χρησιμοποιούν αυτά τα μέτρα. Επίσης η παρότρινση για να ζητούν οι γυναίκες να διεκδικούν θέσεις διευθυντικές, αν υπάρχουν αντίστοιχα μέτρα στο Ευρωπαϊκό, στα Εθνικά Κοινοβούλια και αν βλέπετε και στα δικά σας κοινοβούλια να υπάρχει μια, ε, ένας διαχωρισμός σε σχέση με διαφορετικές μορφές εργασίας και διαφορετικά καθήκοντα στη περίπτωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο, παραδείγματο χάρη, όλοι αυτοί που ασχολούνται με θέματα ασφάλεια είναι άντρε. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω τι απόψει για όλα αυτά τα θέματα. Υπάρχουν ε, κάποιοι ή κάποιες που θέλουν να ζητήσουν το λόγο. Ξεκινάμε με την κυρία Κλειδέτη. Σας παρακαλώ να παρουσιάζετε τον εαυτό σας και να αναφέρετε σε ποιο κοινοβούλιο είσαστε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Λέγομαι τώρα Κλειβέτη, είμαι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λίγους μήνες μονάχα είμαι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έρχομαι από τη Ρουμανία και πρωτού γίνω Ευρωβουλευτής. Ήμουνα εθνική βουλευτής για 8 χρόνια στο Ρουμανικό Κοινοβούλιο και με μεγάλη χαρά σήμερα μπορώ να <clears throat> χαιρετήσω και να καλωσορίσω κάποιες από τις πρώην συναδέλφους μου και άτομα με τα οποία έχω εργαστεί στο Ρουμανικό Κοινοβούλιο στην αίθουσα αυτή. Να σας συγχαρώ καταρχήν κύριε Αντζελίλ και κύριε Γκούσταυσον για τη διοργάνωση αυτού του εξόχου σημαντικού γεγονότος που πιστεύω ότι θα παίξει σημαντικό ρόλο για την περαιτέρω ανάπτυξη των ε, θεμάτων που μας απασχολούν και την εξέβρεση λύσεων για τα προβλήματα της ισότητας των φύλων. Και νομίζω ότι αυτά ενισχύονται από την ε, θετική συμβολή των κοινοβουλευτικών από τα κράτη-μέλη. Η συνθήκη της Λισαβόνας έχει δώσει μεγαλύτερα καθήκοντα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μπορέσει να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά συγχρόνως μας έχει δώσει και την απαραίτητη εμπιστοσύνη για να εξετάσουμε και τη δυνατότητα ενός δικτύου για την ισότητα των φύλων, όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω των εκπροσώπων του και ιδίω μέσω της Επιτροπή για την Ισότητα των Φύλων που εκπροσωπείται από τον κύριο Γκούσταυσον θα μπορούν να συμμετέχουν ώστε τα θέματα αυτά να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν με μια ευρωπαϊκή προσέγγιση. Αν εξετάσουμε την κατάσταση σήμερα, μπορούμε να κατανοήσουμε ότι τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι περίπου τα ίδια. Παντού αντιμετωπίσουμε την ίδια μορφή προβλημάτων και είναι προφανές ότι κάθε κράτος έχει φυσικά την αρμοδιότητα να αποφασίσει για την νομοθεσία περί της ισότητας των φύλων. Αλλά η ύπαρξη ορισμένων <clears throat> νομοθετημάτων ευρωπαϊκού χαρακτήρα, οδηγιών και κανονισμών που θα μπορούσαν να ρυθμίσουν καλύτερα κάποια θέματα όπως η συμμετοχή των γυναικών σε υψηλές θέσεις λήψης αποφάσεων ή άλλες ε, θέσεις που είναι θέσεις υψηλής ευθύνης, ώστε να μπορέσει με τον τρόπο αυτό να επιτευχθεί μια βαθμία μεγαλύτερη ισότητα, αυτό θα ήταν για, την, για μένα μια πολύ θετική επιλογή. Έρχομαι στο πρώτο θέμα το οποίο αναφέρατε κυρία Αντζελίδη. Και θέλω να κάνω εδώ ένα σχόλιο σε σχέση με την κατάσταση του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και εδώ περιλαμβάνω και τους κοινοβουλευτικούς συνεργάτες. <clears throat> Από ό,τι ξέρω υπάρχουν πολλές γυναίκες που είναι μεταξύ των συνεργατών των βουλευτών και από τη μία πλευρά εγώ ως γυναίκα ευρωβουλευτής έχω πολύ καλή σχέση με τις ε, συνεργάτιδές μου και είναι ιδιαίτερα συνειδητοποιημένες για τα θέματα ισότητος των φίλων και ως εκ τούτου πιστεύω ότι μπορούμε στο θέμα αυτό να επενέσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. ότι έχουμε ένα παιδικό σταθμό, κάτι το οποίο βοηθάει τις γυναίκες που εργάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην παιδική φροντίδα οι συνεργάτες μου, <clears throat> η βοηθό μου παραδείγματο χάρη, έχει αυτή την διαβεβαίωση ότι μπορεί να εργάζεται ενώ είναι στον παιδικό σταθμό το παιδί τη και την χάνει της πρέπουσα φροντίδα. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια, αλλά για εμά οι γυναίκε είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά. Γιατί όπω είπατε η εξορρόπηση τη οικογένειακή ζωή και τη επαγγελματική ζωή είναι πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα για τι γυναίκε, περισσότερο από ότι είναι για του άντρε. Θέλω να σταματήσω εδώ Χαίρομαι που μπορώ να συμμετέχω στη σημερινή συνεδρίαση και πάλι θέλω να σας συγχαρώ κύριε Γκούσταυσον και κύριε Αντζελίδη για την πρωτοβουλία αυτής της διοργάνωσης, της θαυμάσιας αυτής της διοργάνωσης. Και θέλω να καλωσορίσω και όλες τις συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ελπίζω θα είναι καρποφόρα συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει συνάδελφος Λάουρισκ, η κυρία Λάουρισκ. Λέγομαι Λάουρεκ Σιμπίλε, είμαι βουλευτής στη Γερμανική Βουλή και πρόεδρος της Επιτροπής για την οικογένεια, τους ηλικιωμένου τις γυναίκες και την νεολαία. Έχω μακρά εμπειρία και από την τοπική αυτοδιοίκηση και ως δικηγόρος στο γραφείο μου ε, και μόνη μου ε, Ανέθρεψα και τα τρία μου παιδιά. Ε, θεωρώ πάρα πολύ σκόπιμο την ευκαιρία που έχουμε σήμερα να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις από πολύ διαφορετικές σκοπιές. Η πολιτική ισότητα, πιστεύω, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, στο μεταξύ έχει φτάσει σε ένα σημείο, και αυτό το βλέπω από τη συζήτηση που παρακολουθώ στη Γερμανία, ένα σημείο λέγω που θα πρέπει να ασχοληθεί με μια βασική έννοια. Γιατί οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται ακόμα σε υψηλά αξιώματα που ασκούν επιρροή. Αυτό είναι το βασικό. Λιγότερο το θέμα της ισότητας, αλλά η επιθυμία των γυναικών να συμμετέχουν στην εξουσία την ίδια και να φτάσουν και σε ένα επίπεδο, να επιθυμούν να φτάσουν σε ένα επίπεδο που επηρεάζει τα πράγματα. Κατά την άποψή μου στην πολιτική ισότητα αυτό δεν έχει συζητηθεί, δεν έχει απασχολήσει ως έννοια. Γι' αυτό δράτω με τις ευκαιρίες για να το αναφέρω έτσι, ε, με τέτοια σαφήνεια. Στη Γερμανία έχουμε πάρα πολλές διατάξεις, νομοθετικές ρυθμίσεις ε, και στη διοίκηση για την ανέλυξη και την ε, επαγγελματική σταδιοδρομία των γυναικών. Για αυτά τα θέματα επίσης έχουμε και πάρα πολλές εκθέσεις που τα τακμηριώνουν. Στη δική μου επιτροπή, στη Γερμανική Βουλή, ασχολούμαστε και αξιολογούμε και τα αποτελέσματα των εκθέσεων και ε, τα συμπεράσματά τους. Και διαπιστώνουμε λοιπόν ότι στα επίπεδα εξουσίας και άσκησης επιρροής ουσιαστικά οι γυναίκες πραγματικά υποεκπροσωπούνται. Έχουν λιγότερη πρόσβαση, αυτό είναι γεγονός. Γι' αυτό εξακολουθεί να τίθεται το αίτημα σε πολιτικό επίπεδο να έχουμε μεγαλύτερη εκπροσώπηση στη διοίκηση ε, της Bundestag. έχουμε πολλές γενικές γραμματείς, ας πούμε και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, δηλαδή όχι ε, το πολιτικό επίπεδο, αλλά ε, στην ε, κεφαλή της διοίκησης και στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Γενικός Γραμματέας, ο Διοικητικός Υπάλληλος είναι γυναίκα. Είναι και άλλα τα Υπουργεία, δεν θέλω να τα παριθμίσω, αλλά αυτά είναι ενθαρρυντικά και μας χαροποιούν και στα μεσαία διοικητικά επίπεδα τα στελέχη είναι πολύ περισσότερα οι γυναίκες από ό,τι στα ανώτατα. Ε, έχετε δίκιο κύριε Αντζελίλη για αυτή τη κρυστάλλινη οροφή που αναφέρετε. Έχει σημασία αυτό διότι οι γυναίκες όταν σχεδιάζουν τη σταδιοδρομία τους δεν λαμβάνουν υπόψη, δεν εκφράζουν από νωρί την επιθυμία να φτάσουν και στα ανώτατα αξιώματα. Τη εξουσία. Νομίζω οι άνδρες όταν προγραμματίζουν την καριέρα τους το σκέφτονται πολύ περισσότερο. Οπότε και σε σχέση με αυτό και με την ιδιωτική οικονομία και τα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων γίνεται μια συζήτηση στη Γερμανία για ποσοστώσεις. Είναι πάρα πολύ επίμαχη και ως βουλευτές έχουμε περιορισμένη βέβαια δυνατότητα επιρροής, αλλά εκεί που μπορούμε ε, θέλουμε να ενθαρρύνουμε τις γυναίκες, να τις προωθούμε και να τις παροτρύνουμε να προετοιμάζονται και για ηγετικές θέσεις. Όπως και εσείς ε, είπατε, διαπιστώνω και εγώ ότι ας πούμε στη χρηματοοικονομία, στη χρηματοπιστωτικά, στις ε, πολύ ψηλέ θέσει δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου γυναίκε. Ε, στη Γερμανία, βέβαια, Έχουμε γυναίκα καγκελάριο που είναι πάρα πολύ γνωστή και πάρα πολύ προβεβλημένη, οπότε μπορεί να συνιστά και ένα πρότυπο για γυναίκες ε, και ένα παράδειγμα και μία απόδειξη ότι μπορούν οι γυναίκες και μπορούν να φτάσουν και σε αυτά τα αξιώματα και να τα καταφέρουν. Ευχαριστώ. Προς το παρόν σταματώ εδώ. Η Πρόεδρος. Σίγουρα η καγκελάριος Μέρκελ μεταξύ άλλων είναι από τις ελάχιστες γυναίκες Πρωθυπουργού. Ωστόσο, ακριβώς δεν πιστεύω ότι ε, είναι και ακριβώς ε, παράδειγμα ε, ανίσχυρης γυναίκας. Επόμενος ομιλητής, Μορέιρα. Ευχαριστώ πολύ. και εγώ θέλω να σας ε, συγχαρώ για την εκδήλωση αυτή που έχετε διοργανώσει. Θέλω να θέσω εντάχει δύο ερωτήματα. Σε σχέση με τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία μπορούν να αναλυφθούν μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή σε ένα Εθνικό Κοινοβούλιο, εμείς στο Πορτογαλικό Κοινοβούλιο έχουμε ποσοστώσεις. Εγώ πάντα υποστήριξα τις ποσοστώσεις αυτές. Διότι δεν νομίζω ότι οι ποσοστώσεις επηρεάζουν την αξιοκρατία για τις γυναίκες. Αντίθετα, οι γυναίκες οι οποίες μπορούν να επιλεγούν βάσει του συστήματος ποσοστώσεων δεν θα μπορούσαν να επιλεγούν λόγω της διάκρισης που ασκεί, ασκείται σε βάρος των γυναικών. Όταν λοιπόν υπάρχει υποχρέωση μιας ποσόστοσης για τις γυναίκες, επιλέγονται μέσα σε αυτή την ποσόστοση οι πιο άξιες γυναίκες. Ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε λοιπόν αυτό το φράγμα διάκρισης που υπάρχει σε βάρος των γυναικών. Για τα συγκεκριμένα τώρα μέτρα συμφιλίωσης της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής που αναφέρθηκαν προηγουμένως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εγώ δεν βλέπω πώς είναι δυνατό να υπάρχει ένας παραδειγματικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έναντι των Εθνικών Κοινοβουλίων, τη στιγμή που δεν υπάρχει διαφορετικό εργασιακό καθεστώς για τις γυναίκες ε, που βρίσκονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις άλλες θέσεις εργασίες. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι οι πρόνοιες που υπάρχουν στην πορτογαλική νομοθεσία θα πρέπει να διευρυνθούν, να τεθούν σε εφαρμογή ευρύτερα να γίνουν ευρύτερα γνώστες. Νομίζω ότι αυτές οι ρυθμίσεις λοιπόν θα ήταν χρήσιμο να γίνουν γνωστές και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αναφέρομαι παραδείγματος χάρη στην γονική άδεια που στην Πορτογαλία μπορεί να χρησιμοποιηθεί <clears throat> και από τον πατέρα και από τη μητέρα. Έχω επίσης κάποιες αμφιβολίες για τις ποσοστώσεις για τις γυναίκες σε υψηλές θέσεις σε ιδιωτικές εταιρείες, γιατί συγκρούεται εδώ η αρχή της ισότητας με την αρχή της, ποσο... της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Φυσικά, εφόσον δεν υπάρχει μια σαφής διάκριση κατά των γυναικών, σε αυτές τις στιγμές η ανεργία στην Πορτογαλία βρίσκεται στο 18%. Είναι μια δραματική κατάσταση και προφανώ οι γυναίκε είναι αυτέ οι οποίε έχουν θίγει περισσότερο από την ανεργία. Πέραν του θέματο λοιπόν των ποσοστώσεων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το οποίο χρειάζεται να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε είναι συνθήκες ίσων ευκαιριών στον εργασιακό χώρο και εδώ αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το αντιμετωπίσει η Ευρώπη και να επιτύχει την ανάπτυξη ενός διαλόγου μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως των χωρών που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση και χρειάζονται μεγαλύτερη οικονομική υποστήριξη. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί οι οποίες θα πρέπει να συζητούν μονάχα με για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την έξοδο από αυτή την τρομερή κρίση που οδηγεί στο να είναι 28 καινούργιοι άνεργοι στην Πορτογαλία κάθε ώρα, αλλά ιδίως για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά σε καθημερινό επίπεδο. Να ξεπεράσουμε λοιπόν απλώς το διάλογο μεταξύ της Κεντρικής, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Δουνουτού και των χωρών που είναι υπό επιτήρηση και να υπάρξει ένας γενικότερος διάλογος μεταξύ όλων των χωρών της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστώ. Μεταξύ άλλων θα ήταν ε, πολύ ενδιαφέρον να αφιερώσουμε μία διάσκεψη στην απασχόληση, στην εργασία και στην ανεργία που χτυπά τις γυναίκες και κυρίως τις νέες γυναίκες γιατί τα στοιχεία για την απασχόληση των νέων που αφορούν τις γυναίκες είναι στοιχεία που όχι μόνο απλώ είναι ανησυχητικά, είναι δραματικά. Έχουμε καθήκον να δώσουμε απαντήσεις, να δώσουμε προοπτικές, να δώσουμε μια ελπίδα σε αυτές τις νεαρές γυναίκες που περιμένουν εκτός από τα εθνικά τους κοινοβούλια αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κοινοτικά θεσμικά όργανα προοπτικές και συγκεκριμένα πράγματα. Πραγματικά μια ολόκληρη γενιά κινδυνεύει να είναι μια χαμένη γενιά, lost generation, όπως την όρισε και ο πρόεδρος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και αυτό αφορά δυστυχώς κυρίως τις νέες κοπέλες και όχι τους νέους άνδρες. Κάτι ακόμα λοιπόν που πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι ότι δεν μπορεί οι γυναίκες να είναι αυτές που θα πληρώσουν το πιο ψηλότερο κόστος για την κρίση γιατί βρίσκονται σε θέση ανισότητας. Είναι απαράδεκτο κάτι τέτοιο. Η κρίση δηλαδή δεν μπορεί να είναι η αιτιολόγηση, η δικαιολογία για να μειώνεται το επίπεδο, για να μειώνεται η επαγρύπνησή μας όσον αφορά την επιβεβαίωση των δικαιωμάτων της γυναίκας. Το λόγο έχει η, η κυρία Φιλάτοβ. Ευχαριστώ. Λέγομαι Τάρια Φίλατοφ και είμαι από τη Φιλανδική Βουλή. Όταν είδα αυτή την επιστολή, λέω, περίεργη υπόθεση. Δεν κατάλαβα το θέμα καν ε, που καλούμαστε να συζητήσουμε. Είναι πάρα πολύ ασαφές και, και πάρα πολύ γενικό. Ας πούμε, βρεφονιπιακή σταθμή, διάφορα θέματα. Η έλλειψη τους δεν πλήττει μόνο τις γυναίκες που δεν μπορούν να πάνε στη δουλειά τους, πλήττει και τους άνδρες. Εμείς στη Φιλανδία οι γυναίκες δουλεύουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχουμε πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία με αυτά τα θέματα και είχαμε και την ευκαιρία την εμπειρία μας να τη μετατρέψουμε σε χρήσιμα εργαλεία για τη ζωή μας. Κάθε επιχείρηση που απασχολεί πάνω από 30 εργαζομένους είναι υποχρεωμένη να έχει πρόγραμμα ισότητας φύλων ε, και να εξασφαλίζει ότι οι γυναίκες τη χάνουν ίσης μεταχείρισης παντού στην εργασία τους, στις απολαβές τους, στις συνθήκες, τα πάντα. Ε, αντίστοιχα εργαλεία έχουμε και δουλεύουν πάρα πολύ σωστά και στο Κοινοβούλιο. διαπιστώσαμε ότι στο παρελθόν οι άντρες και οι γυναίκες είχαν διακριτά καθήκοντα, αλλά προσπαθήσαμε να τα συγκεράσουμε. Και ένα παράδειγμα είναι οι λεγόμενες θετικές διακρίσεις, όπου υπάρχουν ε, λιγότερες γυναίκες ε, που απασχολούνται σε σχέση με τους άντρες. Ελάβαμε μέτρα για να τερματιστεί αυτή η κατάσταση και να εξισορροπηθεί η σχέση. Επίσης, ε, Υπάρχουν διάφορα τείχη που χωρίζουν τα επαγγέλματα σε ανδρικά και γυναικεία και αυτά φροντίσαμε να τα καταρρύψουμε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν συμφωνήσει κάποιος ε, για ένα πρόγραμμα για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την άρση των διακρίσεων, όλα γίνονται δυνατά. Και η νομοθεσία ακολουθεί για να εξασφαλίσει ότι γίνονται με διαφάνεια και με αποτελεσματικότητα και να εντοπίζουμε τις ε, ανισότητες και τις διακρίσεις. Επίσης, οποιαδήποτε νομοθεσία ε, εγκρίνεται θα πρέπει να εφαρμόζεται και φροντίζουμε να ε, παρακολουθούμε και την υλοποίηση παντού. Έχουμε μια συμφωνία στη Φιλανδία που λέγει ότι ανεξαρτήτως κυβέρνησης ε, θα πρέπει να υπάρχει μια υπηρεσία σε κάποιο Υπουργείο ε, που θα ασχολείται με πάρα πολύ σοβαρό τρόπο με αυτά τα θέματα ισότητας. Γιατί υπάρχουν ακόμα διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στο χώρο εργασίας. Γιατί πολλές φορές υπάρχει μια περίεργη αντίληψη για την ιεραρχία ε, στους χώρους εργασίας. Για να σπάσει αυτή θα πρέπει να βοηθήσουμε τις γυναίκες να μπορούν να ανέρχονται στην κλίμακα της ιεραρχίας. Έχουν βελτιωθεί λοιπόν τα πράγματα με τις δράσεις αυτές και στη δημόσια διοίκηση της χώρας αλλά και στην ιδιωτική οικονομία. Επίσης φροντίσαμε να υπάρχει ίση εκπροσώπηση γυναικών στην τοπική αυτοδιοίκηση σε όλα τα επίπεδα. Από το πιο μικρό χωριό μέχρι τη πιο μεγάλη δομή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γενικά, Πιστεύουμε ότι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα ε, ε, για την προώθηση αυτού του θέματος είναι να συνεργάζονται και στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα οι εργοδότες με τα συνδικάτα των εργαζομένων για να πετύχει αυτή η υπόθεση. Ευχαριστώ. E eh, Σας ευχαριστώ και θα ήθελα να καλωσορίσω τη συνάδελφο Αντιπρόεδρο Ποδηματά που είναι υπεύθυνη στο εσωτερικό του Προεδρείου για την επικοινωνία και που όταν ολοκληρωθεί αυτό το πάνελ θα πάρει το λόγο για το θέμα μας. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Ινκοστάντε. Εγώ θα ήθελα Να ευχαριστήσω τους ομιλητές. Φυσικά μας ε, ε, καλούν τα όσα ακούσαμε. Μας καλούν να, να ζητήσουμε και ευκαιρίες για να συσφίξουμε ακόμα πιο στενές σχέσεις μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωκοινοβουλίου. Πιο συγκεκριμένες δε σχέσεις για ορισμένα ζητήματα, για να καθορίσουμε από κοινού τις ε, δραστηριότητες, τις ενέργειες τις οποίες θα πρέπει να προβούμε και από πολιτικό και επικοινωνιακό και από επικοινωνική άποψη να έχει αυτό το θέμα αντίκτυπο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η δράση μας θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική, πιο άμεση, γιατί διαφορετικά αμφιβάλλω κατά πόσο θα υπάρξει δυνατότητα για επιτευξή αποτελεσμάτων ε, επιγόντως ή, εν περιπτώσει, τόσο γρήγορα όσο θα θέλαμε. Το θέμα των γυναικών είναι ένα θέμα δημοκρατικό, χρειάζεται περισσότερη Ευρώπη και άρα σε αυτή τη φάση θα πρέπει να σκεφτούμε πόσο σημαντικό είναι ο ρόλος των γυναικών στην οικοδόμηση μιας πιο προηγμένης ευρωπαϊκής δημοκρατίας και σε σχέση με την δημοκρατική ε, ε, κρίση. Ε, την, περασμένη, την, την τελευταία της παρέμβαση η πρόεδρος Αντζελίλη αναφέρθηκε στην κρίση μιας ολόκληρης γενιάς. Είναι πραγματικά πολύ καυτό το θέμα αυτό και με το μέλλον μας αυτή τη στιγμή γιατί η κρίση που βαραίνει περισσότερο τις γυναίκες και τους νέους που αναζητούν δουλειά μπλοκάρει και την διαδικασία οικοδόμησης του μέλλοντος ποσοστά αναπαραγωγής και γεννητικότητας που διαρκώς μειώνονται δεν μπορεί παρά να μας ανησυχεί ένα καμένο μέλλον στο οποίο η Ευρώπη δεν μπορεί να μείνει άπρακτη η κρίση ε, είναι όμως ταυτόχρονα μια δημοκρατική και οικονομική ευκαιρία όπου το δυναμικό των γυναικών και από οικονομικής άποψης δεν μπορεί να το ξεχνάμε ή να τα αφήνουμε χρησιμοποιητό, ανεκμετάλλευτο ε, δεδομένε της ε, πολύ μεγάλης παιδείας που έχουν οι γυναίκες και του δυναμικού που έχουν. Εγώ πιστεύω πως θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια για να βελτιώσουμε τους ίδιους τους κανονισμούς του Ευρωκοινοβουλίου και του κανονισμού των Εθνικών Κοινοβουλίων. Αυτό είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να το εξετάσουμε ει βάθο. γιατί στην εκπροσώπηση των επιτροπών και στην κατανομή των αξιωμάτων όλα εξαρτώνται από τη διακριτική ευχαίρεια για τη βούληση των κομμάτων. Εγώ πιστεύω πω θα πρέπει να γίνει ένα ακόμα βήμα μπροστά για να οριστούν κανόνε, να αλλάξουν οι κανονισμοί αυτοί να είναι αυτή μια δέσμευση που μπορούμε να την αναλάβουμε. Σε σχέση με τη συμβιλίωση ε, εργα επαγγελματικής ζωής και οικογενειακής ζωής. Θα πρέπει να γίνουν κάθε είδους προσπάθεια και στο πλαίσιο των οδηγιών και των προγραμμάτων να επιμείνουμε για τη δυνατότητα αναδιοργάνωσης της εργασιακής δομής. Δηλαδή χρειάζεται πέρα από την ε, συμφιλίωση μεγαλύτερη ευελιξία στην οργάνωση της εργασίας για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των γυναικών για τις ποσοστώσεις της επιχειρήσης. Εμείς στην Ιταλία φτιάξαμε μια, ένα νόμο που πέρασε από το Κοινοβούλιο όσον αφορά τις εταιρείε που είναι εισηγμένε στο χρηματιστήριο και εδώ θα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι στην ολόκληρη την Ευρώπη και με βάση την επόμενη οδηγία, αυτό είναι ένα άλλο πεδίο πάνω στο οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε και ίσως και να ε, επιμείνουμε ώστε να προωθηθεί αυτή η οδηγία. Νομοθεσίες που θα προωθούν του μηχανισμούς εκπροσώπησης των γυναικών Επίση. Χρειάζονται δηλαδή πιο συγκεκριμένες νομοθεσίες σε σχέση, βέβαια, ανάλογα με την αυτονομία των χωρών και τα συντάγματά τους. Αλλά πραγματικά διερωτώ δεν μπορεί να κάνει περισσότερα η Ευρώπη για να ορίσει και έναν δείκτη για την παρουσία των γυναικών, έναν δείκτη για, τα, για το φύλλο και να επιφέρει κάτι τέτοιο και κάποιες κυρώσεις όσον αφορά τις σχέσεις. Τα λέω τώρα συνοπτικά, είναι ιδέες αυτές να δώσουμε μεγάλη προσοχή. Δίνουμε μεγάλη προσοχή στα περιβαλλοντικά ζητήματα, ας πούμε. Προτείνουμε μηχανισμούς κυρώσεων. Με τον ίδιο μηχανισμό δεν θα μπορούσαμε και εφόσον αποφασίζουμε ότι είναι ένας παράγοντας δημοκρατικός και οικονομικός για την Ευρώπη, δεν θα μπορούσε να έχει την ίδια σημασία και άρα να μελετήσουμε αντίστοιχους μηχανισμούς. Τελευταίο ερώτημα. Είναι προφανέ ότι ο πρώτο επόμενο αγώνα που θα μα ε, απασχολεί σαν αυτή η οδηγία στην οποία αναφερθήκατε, συγκεκριμένα για την εκπροσώπηση στι ε, τοπικέ ε, στις τοπικές αρχές. Εμείς είμαστε στο Γερουσία αυτή τη στιγμή με ένα νόμο που αφορά τη διπλή προτίμηση και σε σχέση δηλαδή με το Σύνταγμά μα μπορεί κανεί να υποδείξει δύο προτιμήσει. Μία μπορεί να είναι προαιρετική. Αν όμω επιλέξει να κάνει δύο δύο επιλογές, δύο προτιμήσεις θα πρέπει να είναι και διαφορετικού φύλου. Ίσως αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει και ήδη έχει γίνει αυτό ας πούμε, σε μια περιφόρεια, να υπάρξει έτσι μεγαλύτερη εκπροσώπηση. Πιο συγκεκριμένε προτάσεις λοιπόν και κοινέ δράσεις πολύ πιο ισχυρέ. Σας ευχαριστώ. Grazie, eh, Ευχαριστώ κυρία Μανατίδου παρακαλώ. Prego. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι η Αμανατίδο Ευαγγελία, εκπροσωπώ την Ελληνική Βουλή. Είμαι εδώ ως πρώτη αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας ε, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ε, είναι πολύ σημαντική η σημερινή συζήτηση σε επίπεδο κρατών μελών της Ευρώπης. Να μεταφέρω βεβαίως και ένα κλίμα από την Ελλάδα που το τελευταίο διάστημα έχει γίνει και ε, το πρώτο θέμα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε παγκόσμιο επίπεδο ε, για αυτό που συζητούμε, σας άκουσα κυρία Αντελήλη και κύριε Γκούσταυσον και συμφωνώ σε αρκετά από αυτά όπως έχω διαβάσει και τις εκθέσεις ε, που ε, μας έχουν δοθεί για αυτήν την συνάντηση σήμερα. Έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Θέλω να σας μεταφέρω εγώ τα δικά μας ποσοστά από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, διότι ε, ε, θα ήθελα να μιλήσω στην επόμενη, όπως και θα μιλήσω για το γυναίκα και πολιτική, αλλά εμπλέκονται όλα αυτά τα θέματα μεταξύ τους, οπότε μπορεί κάποια πράγματα να τα πω και τώρα. Εμείς στην ε, ε, στο προσωπικό της ε, Βουλής των Ελλήνων ε, έχουμε υψηλά ποσοστά γυναικών. Το ποσοστό γυναικών εκεί είναι 57% και των ανδρών είναι 43%. Το ποσοστό των γυναικών σε υψηλόβαθμες θέσεις είναι 54% έναντι 46% των ανδρών. Αυτό όμως ισχύει μόνο για το προσωπικό μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Έξω η αντιστοιχία δεν είναι αυτή. Όπως επίσης και έχουμε ένα ποσοστό σε επίπεδο ελληνικής βουλής γυναικείας εκπροσώπησης 63 γυναικών βουλευτών ε, δηλαδή το, στους 300, δηλαδή 21%. Βέβαια είμαστε μακριά από το ποσοστό του 6,3 που υπήρχε το 1996 στην Ελληνική Βουλή. Ε, άρα μπορούμε να πούμε ότι πηγαίνουμε σε μια καλύτερη εκπροσώπηση αν και είναι από τις χαμηλές ακούγοντας και τον μέσο όρο που ε, θέσατε σε επίπεδο ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα ε, εμείς έχουμε θεσμοθετήσει το 1 τρίτο ε, του φύλου ε, ως ποσόστοση στις, και στις εθνικές αλλά και στις αυτοδιοικητικές εκλογές στις, στους Δήμους δηλαδή και στις 13 περιφέρειες των, της χώρας μας αλλά από εκεί και πέρα ε, δεν είναι μόνο, και το είπατε με έναν τρόπο κυρία Τζελίλη ε, δεν είναι η, τη γυναίκα να βάλουμε ποσόστοση, είναι να, ε, υπάρχει, να υπάρχουν οι δυνατότητες, οι δομές, η γυναίκα από μόνη της να μπορέσει να μπει στα κέντρα λήψη των αποφάσεων, πιο μπροστά να έχει ασχοληθεί βεβαίως με την πολιτική, αυτή μπορεί να είναι και συνδικαλισμό στον εργασιακό της χώρο, ε, αλλά ε, στην Ελλάδα έχουμε ε, μία, γι' αυτό ξεκίνησα και από την αναντιστοιχία, έχουμε ελάχιστες δομές που βοηθούν, ειδικά σήμερα στην οικονομική κρίση, την Ελληνίδα να ασχοληθεί με θέματα όπως είναι η πολιτική και ο συνδικαλισμός διότι και η παιδεία αλλά και οι κοινωνικές δομές που θα βοηθήσουν την εξέλιξη της Ελληνίδας και ε, στον εργασιακό χώρο και στην εκπαίδευσή της ακόμη είναι σε χαμηλά επίπεδα. Ε, την ώρα που κόβουν η ανεργία των γυναικών και ειδικά των νέων είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, την ώρα που η ανασφάλιστη εργασία ειδικά στις γυναίκες και στους νέους είναι επίσης σε πολύ υψηλά επίπεδα, την ώρα που υπάρχει εργοδοτική τρομοκρατία ειδικά στις γυναίκες και θα σας θυμίσω ε, ένα γεγονός που είχε κάνει το γύρο του κόσμου και ήταν η Κούνεβα ήταν η Βουλγάρα που ε, τη συμπεριφέρθηκαν με αυτόν τον τρόπο η συνδικαλίστρια καταλαβαίνετε ότι στην Ελλάδα είναι διαφορετικά τα στοιχεία από αυτά που αρχικά σας, ε, παράθεσα. Ε, το θέμα είναι το πώς μπορεί να στηριχθεί ε, η ισότητα των φύλων γιατί ε, σίγουρα είναι η ίση ε, εργασία και η ίση αμοιβή για την ίδια εργασία είναι το σημαντικότερο από όλα αλλά τώρα ζούμε στη χώρα μας μέσα από, από τα μνημόνια και τα μέτρα, τα νέα μέτρα που περιμένουμε σκληρές συνθήκες διαβίωσης και ειδικά όπως είπα και για τις ε, ε γυναίκες κλείνουν παιδική σταθμή άρα εδώ είναι ένα ακόμη πλήγμα ε, για τον γυναικείο πληθυσμό ε, κλείνουν κοινωνικές δομές αυτές οι ελάχιστες ε, υποχρηματοδοτούνται το βοήθεια στο σπίτι που είναι δομή για τα άτομα με αναπηρία για τους ηλικιωμένους άρα επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο η γυναίκα με όλα τα υπόλοιπα συν αυτά και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό για να, ε, γιατί τελειώνει και ο χρόνος μου, είναι πολύ σημαντικό να δούμε την γυναίκα μέσα στην ε, κρίση, να βοηθηθεί την, και την άσκηση βεβαίως της ε, πολιτικής από γυναίκες που είναι πάρα πολύ σημαντική και θα πρέπει αυτή να διακατέχεται από ευαισθησία και από κοινωνική δικαιοσύνη γιατί σίγουρα η γυναίκα έχει άλλα αισθητήρια χωρίς να θέλω να προσβάλλω τους άνδρες ε, που παρευρίσκονται ε, στην σημερινή συζήτηση και ειδικά τον κύριο Γκούσταυσον ο οποίος είναι και ο πρόεδρος της Επιτροπής ε, αλλά θα πρέπει να υπάρχει πάντα ε, εκείνη η γυναικεία διέστηση στην άσκηση της πολιτικής διότι αλλιώς θα είμαστε ένα κακό κακέκτυπο ε, του αντρικού προτύπου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Έχουμε ακόμα δύο παρεμβάσεις. Θα δώσουμε ακόμα σε δύο μιλητές ε, το λόγο. Κυρία Τόμα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την οργάνωση αυτής της εκδήλωσης σήμερα. Θα ήθελα να παρουσιάσω την κατάσταση της Εστονίας. Έχουμε 101 βουλευτές στο Εστονικό Κοινοβούλιο, 19 από τους οποίους είναι οι γυναίκες, περίπου ένα πέμπτο. Έχουμε συζητήσει το θέμα των ποσοστώσεων κατ' επανάληψη και στα μέσα ενημέρωσης και στον πολιτικό στίβο και υπάρχει μεγάλη, ε, μεγάλη επιφυλακτικότητα γιατί στην Πορτογαλία όπως αναφέρθηκε υπάρχουν ποσοστώσεις αλλά δεν λειτουργούν. Το ερώτημα είναι κατά πόσο θα πρέπει να επιφέρουμε και τις ποσοστώσεις για δουλειές χαμηλών αμοιβών, ώστε να υπάρχουν και πιο πολλοί άνδρες οι οποίοι αναλαμβάνουν τις εργασίες αυτές χαμηλών αμοιβών. Τα έχω παρακολουθήσει όλα αυτά πολύ προσεκτικά, αλλά είμαι μητέρα πέντε παιδιών, είμαι βουλευτής και προσωπικά δεν αντιμετώπισα δυσκολίες. Αλλά ίσως ήμουν απλώς τυχερή. Αν δείτε όμως γύρω σας, δεν ξέρω Πόσοι άντρες είναι σήμερα σε αυτή την αίθουσα. Λιγότερο από 10%. Πιστεύω ότι η ισότητα των φίλων είναι αυτή τη στιγμή ένα θέμα καθαρά γυναικείο. Οι άντρες δεν ενδιαφέρονται. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Γκούσταυσον. Γιατί γίνεται αυτό. Γιατί παραγωγικά στην κοινωνία μας έχουμε μια τέτοια κατάσταση. Από τις 19 γυναίκες στο Ιστορικό Κοινοβούλιο οι μισές είναι χωρισμένες. Γιατί σε τελική ανάλυση οι άνδρες είναι που δημιουργούν αυτή την, όπως αναφέρατε, κρυστάλλινη οροφή. Οι γυναίκες οι οποίες είναι παντρεμένες θα πρέπει να κάνουν μια επιλογή. Η οικογένειά τους ή ο χώρος εργασίας. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ ωραίο να τα συζητάμε μεταξύ μας. Είναι πολύ θετικό ότι γίνεται αυτή η συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το μήνυμα όμως κάποτε θα πρέπει να φτάσει και τους άντρες. Να μεταφράσετε σε μια γλώσσα που καταλαβαίνουν και οι άντρες. Δεν ξέρω αν αυτό είναι η υπόθεση των μέσων ενημέρωσης ή κάποια άλλοι. Πρέπει να ξεπεράσουμε τα στερεότυπα. Ό,τι ποσοστώσεις και να εφαρμόσουμε, τελικά χρειάζεται μια επιλογή. Ο άντρα μου μου είπε, ή πήγαινε στην πολιτική ή να ασχολείσαι με την οικογένειά σου και ξέρετε ποια επιλογή έκανα εγώ. Ε, ε, Ευχαριστώ. Τελευταία, τελευταία παρέμβαση σε αυτό το πάνελ. Οκτεν. Και εγώ θέλω να σας συγχαρώ για την διοργάνωση αυτής της μεγάλης και τόσο σημαντικής ε, διοργάνωσης Θα ήθελα να αναφερθώ στην ε, κατάσταση της ε, Τουρκίας και τα ενισότητα των ε, φύλων. Η Τουρκία έχει κάνει κάποιες συνταγματικές πρόνοιες για να εξασφαλίσει την ισότητα των ανδρών και των γυναικών. Στη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση έχει δημιουργηθεί η Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών για τις Γυναίκες που ενεκρίθη η δημιουργία της στις 25 Φεβρουαρίου 2009 και θεσπίστηκε στις 25 Μαρτίου 2009. Η Επιτροπή αυτή είναι αρμόδια για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και της πρόθεσης των δικαιωμάτων αυτών και της ισότητας ανθρώπων και γυναικών. Εκπροσωπούνται τα κόμματα σε αυτή την Επιτροπή επί τη βάση αριθμητικής τους δύναμης και η Επιτροπή μας είναι μία από τις λίγες επιτροπές η οποία περιλαμβάνει και ανεξάρτητους βουλευτές. Όπως θα μπορούσατε να φανταστείτε, τα περισσότερα μέλη αυτής της Επιτροπής είναι ε, γυναίκες. Στην προηγούμενη θητεία 11 από 17 ήταν γυναίκες. Στην τωρινή θητεία 20 από 26 είναι γυναίκες. και όλο και περισσότερο αυξάνει η συμμετοχή γυναικών σε αυτή την επιτροπή. Επίσης, η συμμετοχή στο, στη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση των Γυναικών έχει αυξηθεί σημαντικά. Από 4,4% το 2002 έχει φτάσει στο 9,1% το 2007 με 48 βουλευτές γυναίκες και είναι τώρα 14,1% με 78 γυναίκες στη Βουλή που εξελέγει το 2011. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική πρόοδος για την επίτευξη της ε, ισότητας ανδρών και γυναικών που θέλουμε να επιτευχθεί το 2015 όπως αναφέρεται στην έκθεση για τους στόχους της χιλιετίας. στο τουρκικό κοινοβούλιο τα παιδιά του προσωπικού που είναι μέχρι 6 χρονών έχουν πρόσβαση στον παιδικό σταθμό. Έχουμε λοιπόν 100, ε, περίπου 500 γυναίκες συνολικά που εργάζονται στο κοινοβούλιο και είναι 35% του συνολικού προσωπικού. Μέσα στην προσπάθεια επίτευξης ισότητα των φύλων σε διεθνέ επίπεδο, η Τουρκία έχει συμβάλει στην εκπόνηση τη σύμβαση του Συμβουλίου τη Ευρώπη για την καταπολέμηση τη βία κατά των γυναικών και τη βία στον οικιακό χώρο. Και κατά την Προεδρία της Επιτροπής των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης το 2011, η Τουρκία συνέβαλε ιδιαίτερα στο θέμα αυτό και υπέβαλε τις ε, προτάσεις της στην Επιτροπή αυτή το Μάρτιο του 2011 ε, και από το 2012 η Τουρκία είναι η πρώτη χώρα η οποία έχει κυρώσει την σύμβαση αυτή για τη βία κατά των γυναικών. Βάση. Επίσης έχει προωθήσει ένα κοινό πρόγραμμα για την ισότητα των φύλων στην Τουρκία. Αυτό είναι το μεγαλύτερο σχέδιο στο οποίο έχει εμπλακεί η Επιτροπή μας μέχρι τώρα, μαζί με τις, ε, το πρόγραμμα ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Μέσα στα πλαίσια αυτού του σχεδίου που έχει διάρκεια δύο ετών έχουν λάβει χώρα και θα λάβουν χώρα περαιτέρω ενέργειες σε εθνικό και τοπικό επίπεδο για να γίνουν ευρύτερα γνωστές οι πολιτικές ισότητε των φύλων της τουρκικής δημοκρατίας και να υπάρξει και μεγαλύτερη συνειδητοποίηση του κοινού για τα θέματα αυτά. Αυτές οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν μέτρα ευαισθητοποίησης ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ισότητα στον κοινωνικό χώρο μεταξύ ανδρών και γυναικών. Μέσα στα πλαίσια λοιπόν αυτού του σχεδίου έλαβαν χώρα συναντήσεις και με εκπροσώπους των τοπικών ε, υπευθύνων, των ε, ε, διοικητών των, των νομαρχών και των άλλων αρχών, ώστε να μπορέσει να προωθηθεί η ισότητα σε κάθε περιοχή. Και μετά από το πρωτόκολλο το οποίο υπεγράφει με τις τηλεπικοινωνιακές αρχές της Τουρκίας, υπήρξε και η εκτύπωση σε, μπροσούρ, μπροσούρες που ε, υποστηρίζουν την ισότητα των φύλων και καταδικάζουν τη βία κατά των γυναικών. Όλες αυτές οι μπροσούρες έχουν διανεμηθεί σε κάθε νοικοκυριό στην Τουρκία. Και επίσης έχουν εκδοθεί γραμματόσημα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στο ταχυδρομείο και υποστηρίζουν ακριβώς αυτές τις ενέργειες. Ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστώ. Έχουμε κάπως αργήσει. Οπότε ζητώ συγγνώμη από τους συναδελφούς ε, Ποδηματά και Κάρας, αλλά η συζήτηση ήταν πραγματικά ενδιαφέρουσα. Πριν να δώσω το λόγο στους συναδέλφους όμως, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην, ε, στον πρόεδρο Γκούσταυσον, διότι το, η κυρία Τούμα τον ρώτησε κάτι συγκεκριμένο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να απαντήσω ναι. Ανέφερα στην πρωτομιλία μου τη χρηματοοικονομική κρίση και τις επιπτώσεις που έχει, τις διαφορετικές στους άνδρες και τις γυναίκες. Αναφερθήκατε και πολλοί από εσάς αυτό το θέμα. Σε σχέση με αυτό, επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω το εξής. Η κρίση πλήττει με διαφορετικό τρόπο άνδρες και γυναίκες, αλλά οι γυναίκες δεν θα πρέπει να θεωρούνται πάντα μόνο θύματα ε, της κρίσης, αλλά και ένα τμήμα της λύσης. Γι' αυτό στις 8 Μαρτίου του 2013 ε, θα διοργανώσουμε μία ε, διάσκεψη με θέμα η απάντηση των γυναικών στην κρίση, επευκαιρία της 8ης Μαρτίου. Γιατί εμείς δεν θεωρούμε ότι μέχρι τις 8 Μαρτίου θα έχει τελειώσει η κρίση. Αν έχει τελειώσει, μπράβο, να χαρούμε. Αλλά νομίζω ότι και τότε θα είναι επίκαιρο αυτό το θέμα. Ένα άλλο ερώτημα που μου έθεσε η κυρία το Απαντώ σύντομα. Κανονικά θα ήθελα πολύ περισσότερο χρόνο για να το αναλύσω πάνω από ένα δίλεπτο. Με ρωτήσατε για ποιο λόγο η ισότητα συχνά θεωρείται ζήτημα γυναικείο και παραμένει. Ναι, και εγώ αναρωτιέμαι. Κοιτάξτε ποιος είναι ο λόγος. Η, κοινωνία μας δεν είναι κοινωνία ισότητας. Ζούμε σε μια κοινωνία που κατά την άποψή μου έχει μια ε, οργάνωση εξουσίας και είναι η διαφορετική εξουσία των ανδρών και των γυναικών και για να είμαστε ειλικρινεί, οι γυναίκες έχουν λιγότερες εξουσίε. Γενικά υπάρχουν και εξαιρέσει, βέβαια, ε, αλλά μπορεί κανείς αυτό να το χαρακτηρίσει πατριαρχική κοινωνία ή εγώ το λέω κοινωνία διεράρχηση ε, των φίλων, εν πάση περιπτώσει. Έτσι έχουν τα πράγματα, είναι πατριαρχική η κοινωνία μας, γι' αυτό ε, έχουμε αυτή τη συζήτηση και στερεότυπα και ρόλους γυναικείους, ανδρικούς, από μικρούς έτσι μας μεγαλώνουν. Με τέτοια στερεότυπα από τα γενοφάσκια μας θα πρέπει να απελευθερωθούμε από αυτά τα ε, στερεότυπα. Ε, είναι κοινωνική λοιπόν αυτή η αιτία και δεν είναι καθόλου βιολογική. Και πού οδηγεί αυτό η συμπεριφορά μας φαίνεται στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η κοινωνία ίδια. Γίνεται λόγος για τη σημασία ε, της υγείας, ε, της ε, φροντίδας των παιδιών, για να μπορούν, λέει, σε αυτά τα επαγγέλματα να εργάζονται γυναίκες. Όπως είπε όμως και κάποιος προηγουμένως, το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για τους άνδρες. Αλλά φαίνεται δεν το βλέπει κανείς έτσι. Διότι όταν προάγεται ένα άνδρας ή ε, ανεβαίνει στην ιεραρχία, δεν τον ρωτάει κανείς και τώρα τα παιδιά σου τι θα τα κάνεις. Όταν προάγεται μια γυναίκα όμω και ανεβαίνει τα κλιμάκια, τη ρωτάνε και την οικογένειά σου τι θα την κάνεις. Ε, για μένα το θέμα της ισότητας δεν είναι θέμα γυναικείο καθόλου, είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατία. και θα πρέπει αυτό να είναι ευθύνη όλων. Διότι σε όλα τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, συμμετέχουν οι άνδρες με τρόπο πάρα πολύ δραστήριο. Αυτή τη στιγμή γίνονται αυτά θέματα ισότητας, εξαφανίζονται οι άνδρες ε, ως διαμαγείας. Ε, και πραγματικά είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όχι γυναικείο ζήτημα. Έτσι, απαντώ στην ερώτησή σας. Bene. Μάλιστα. Μια τελευταία πληροφορία που ήθελα να σας δώσω σε σχέση ε, με τις γυναίκες ευρωβουλευτές του Ευρωκοινοβουλίου είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι παρότι είναι οι εικόνες του Κοινοβουλίου είναι σε σχέση με την ε, δραστηριότητα, την κοινοβουλευτική πολύ δραστήριες. Εγώ ε, για την Ιταλική αντιπροσωπία την οποία γνωρίζω καλύτερα να σας πω ότι είμαι ευτυχής και περήφανη που μπορώ να σας πω ότι οι γυναίκες της αντιπροσωπείας μου είναι αυτές οι οποίες είναι πολύ εφοσιωμένε ε, τόσο όσον αφορά την παρουσία του στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι πραγματικά υποδειγματική η συμπεριφορά τους, ακόμα και όταν ε, τιμωρούνται εντό ε, εισαγωγικών, αυτό δεν τι αποθαρρύνει. Αντίθετα, δουλεύουν ακόμη περισσότερο. δώσω το λόγο στους δύο συναδέλφους, την κυρία Ποδηματά και τον κύριο Κάρας, που είναι υπεύθυνοι για την επικοινωνία, υπογραμμίζοντας απλά ότι από πλευράς όλων εκτιμήθηκε αυτός ο στόχος ε, δικτύωσης, ανταλλαγής πληροφοριών, καλών πρακτικών, την, η ενημέρωση ήδη είναι συμμετοχή δυνατότητα να ενημερώνονται οι πολίτες, να συμμετέχουν, να εμπλέκονται, να μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, πράγματα για τα οποία χρειαζόμαστε οπωσδήποτε αυτή τη στιγμή. Uh, Ευχαριστώ, Ρομπέρτα. Ευχαριστώ, Αντιπρόεδρε Αντζελίλη. Και για την ευκαιρία που μου δίνετε ε, να βρίσκομαι εδώ σήμερα ανάμεσά σας η μαζική συμμετοχή στη διάσκεψη αυτή, όσο και η ποιότητα των παρεμβάσεων που είχα την ευκαιρία να ακούσω, αποδεικνύουν ότι η πρωτοβουλία πάντα στέφεται με επιτυχία. Αλλά ε, είναι και μια ακόμα απόδειξη της πολύτιμης συνεισφοράς των γυναικών στην πολιτική. Επιτρέψτε μου καταρχάς να σας συγχαρώ λοιπόν και σας ε, προσωπικά και τον πρόεδρο της Επιτροπής Γυναικών, τον κύριο Κούστευσον, για την πρωτοβουλία αυτή να συναντήσουμε τους ομολόγους μας των Εθνικών Κοινοβουλίων και να έχουμε σε βάθος ανταλλαγή απόψεων για την ισότητα των φύλων. Η Ευρώπη ζει κρίσιμες στιγμές για την ολοκλήρωσή της, για το μέλλον της, για το ευρωπαϊκό εγχείρημα το ίδιο. Και πιστεύουμε ότι η πλήρη συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων και ενίσχυση και σύσφυξη των δεσμών και των σχέσεών μας είναι προϋπόθεση επιτυχίας. Και αυτό σίγουρα έχει να κάνει και με θέματα ισότητας των φύλων. Θα ήθελα λοιπόν να αποτίσω ένα ιδιαίτερο φόρο τιμή στην επιμονή ε, της Προέδρου Αντζελίλη, της Αντιπροέδρου του Κοινοβουλίου, που έκανε δυνατή αυτή την ε, συνάντηση. Είναι ευκαιρία λοιπόν όχι μόνο να ανταλλάξουμε πρακτικές, αλλά και να τονίσουμε ότι παρά τις πρόοδους που έχουν γίνει στην ισότητα των φύλων, απομένει ακόμα πάρα πολλή δουλειά και πολλής δρόμος να διανύσουμε. Ο Αντιπρόεδρος Κάρας και εγώ προσωπικά χαιρόμαστε που έχουμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε πλήρως ως αρμόδια αντιπρόεδροι για θέματα επικοινωνίας και πληροφόρησης, διότι πιστεύουμε ότι κάθε δράση του Κοινοβουλίου θα πρέπει να διαβιβάζεται στους πολίτες, να είμαστε κοντά στους πολίτες. Αυτό σημαίνει να εργαζόμαστε προς όφελός τους, για να βελτιώνονται οι ζωές τους. Να μαθαίνουν οι πολίτες τι κάνουμε εμείς ε, για εκείνους, αλλά να μαθαίνουμε και από εκείνους τι γίνεται. Δηλαδή αυτή η οδός επικοινωνίας είναι διπλής κατεύθυνσης. Εμεί λοιπόν οι δύο αντιπρόεδροι που έχουμε αυτή την ευθύνη θα προσπαθούμε να τονίζουμε κυρίως τις προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επικοινωνεί και να προωθεί το θέμα της σώτας των φύλων. Και ένα παράδειγμα είναι και η σημερινή συνεδρίαση, η σημερινή διάσκεψη για την προώθηση των φύλων. Με την υποστήριξη των ε, αρμοδίων υπηρεσιών του Κοινοβουλίου ε, στέλνουμε σήμερα ένα μήνυμα σε όλη την Ευρώπη από τα γραφεία πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη-μέλη, από τους αρμοδίους προσώπους τύπου, από την ιστοσελίδα του κοινοβολείο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλες επιγραμμικές ε, πλατφόρμες. Όπως γνωρίζετε μεταδίδεται απευθεία στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή η συνεδρίαση και μπορούν να παρακολουθούν ε, όσοι πολίτες ενδιαφέρονται τη διοργάνωση αυτή. Χτες προπαρασκευαστικά είχαμε ένα σεμινάριο για δημοσιογράφους όπου εξετάστηκε σε βάθος η ισότητα των φύλων για να έχουν τα απαραίτητα εφόδια και τη γνώση οι δημοσιογράφοι να εμβαθύνουν σε αυτό το θέμα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αφουσιωμένο στο θέμα της ισότητας των φύλων ε, και ε, κάνει πολλές ε, τέτοιες δραστηριότητε με αποκορύφωμα την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Όπως γνωρίζετε την 8η Μαρτίου κάθε χρόνο γιορτάζουμε τα επιτεύγματα των γυναικών, τα παρελθόντα, τα σημερινά και τα μελλοντικά σε διάφορους τομείς της κοινωνίας. Κάθε χρόνο και στο Κοινοβούλιο ε, υπάρχει ένα θέμα που επιλέγουμε και μάλιστα το επιλέγει η Επιτροπή Γυναικών και Ισότητας Φίλων το Νοέμβριο. Φέτος ακούσαμε από τον πρόεδρο της Επιτροπής Γυναικών πριν από λίγα λεπτά ε, το πάρα πολύ ε, εύστοχο και επίκαιρο θέμα που θα επιλέξουν για φέτος. Το 2012 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργάνωσε τρεις μεγάλες εκδηλώσεις στις Βρυξέλλες με θέμα ε, τις ίσες αμοιβέ. Διότι όπως γνωρίζετε το 2012 είχε ως έμβλημα ίση αμοιβή για ε, εργασία ίσης αξίας. Επίσης και στα κρατημέλη, στα κατατόπους γραφεία κάναμε εκδηλώσει. Θα πρέπει να στείλουμε το μήνυμά μας εκτός των τυχών του Κοινοβουλίου και εκτός Βρυξελών. Να φτάσουμε κοντά στους πολίτες, όπου αυτοί και αν βρίσκονται. Να ενισχύουμε τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την αφοσίωσή του ε, σε αυτά τα θέματα της ισότητας, αλλά επιτόπου, κοντά στους πολίτες. Για να φτάσουμε σε αυτό λοιπόν το στόχο θα πρέπει να είναι η επικοινωνία αμφίδρομη, για να ε, μαθαίνουμε κι εμείς τι λέγουν οι πολίτες, ποιες είναι οι εμπειρίες τους, οι ανάγκες τους, τι ζητούν από μας ε, και ε, πώς βρίσκουν τις δράσεις μας όλα τα μέσα αξιοποιούνται, τα κοινωνικά μέσα και οι διάφορες πλατφόρμες και σήμερα έχουμε πολύ περισσότερες ευκαιρίες από ό,τι στο παρελθόν για να έχουμε ένα γνήσιο και συγκεκριμένο διάλογο με τους πολίτες. Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε όλα τα νέα μέσα χωρίς να εγκαταλείπουμε τις ε, παραδοσιακές μεθόδους επικοινωνίας και πληροφόρησης. Ωστόσο, εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε ακόμα παραπέρα από την επικοινωνία αυτή με μονομένα θεματικά ε, γεγονότα και δράσεις, μια καμπάνια να έχουμε για τα θεμελιώδη δικαιώματα που ε, πρεσβεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και όπως είπε προηγουμένως και ο κύριος Γκούσταυσον, η ισότητα των φύλων είναι ένα τμήμα των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μια κληρονομιά πολιτικών αποφάσεων και ε, νομοθετημάτων και χωρίς καμιά αμφιβολία είναι υπέρ της δημοκρατίας, ελευθερίας, της έκφρασης, ε, υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της πολιτιστικής πολυφωνίας με ευρεία πολιτική συνένεση σε αυτές τις ε, κομβικές και βασικές αξίες. Σήμερα ζούμε μια πολύ πλευρή ε, κρίση και πολύ επίπεδη και μεταξύ αυτών και κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών για τα θεσμικά τους όργανα και οι αξίες ε, προάγουν και ε, προωθούν το βασικό και εκτιμένο. Οι πολίτες πρέπει να είναι περήφανοι που συμμετέχουν σε μια ένωση που γίνεται βαθύτατα σεβαστό το θέμα των αξιών. Ωστόσο, δεν είναι στο κενό οι αξίες. Μεταφράζονται σε νομοθεσία, σε νομοθετική δουλειά, σε συγκεκριμένες πολιτικές, σε τομείς που ε, άπτονται άμεσα της καθημερινής ζωής των πολιτών. Όταν λοιπόν επικοινωνούμε για θέματα ισότητας των φύλων δεν είναι κάτι γενικό και αόριστο, αλλά εστιάζουμε στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη σχετική νομοθεσία καθ' όλη τη διάρκεια της νομοθετικής ε, δραστηριότητας. Τέλος, θέλω να απευθύνω μια έκκληση σε όλους εμάς που εκπροσωπούμε τους πολίτες της Ένωσης. Νομίζω ότι αυτό που χρειαζόμαστε, αυτό που πρέπει να κάνουμε, να ακούμε περισσότερο τους πολίτες. Πρέπει να σας ενημερώσω ότι σύμφωνα με το τελευταίο ευρωβαρόμετρο, που γνωρίζετε ότι είναι η δημοσκόπηση στην Ευρώπη της κοινή γνώμης, οι βασικές αρχές που θα πρέπει να προωθεί και να υπερασπίζει το Κοινοβούλιο είναι τα εξή. Πρώτον, προστασία ανθρωπίνων των δικαιωμάτων Δεύτερον, ισότητα ανδρών και γυναικών, ελευθερία έκφρασης, τρίτον, τέταρτον, αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών, αλληλεγγύη μεταξύ της Ευρώπης και των φτωχότερων κρατών του κόσμου. Προστασία μειονοτήτων, προώθηση πολυπολιτισμικού διαλόγου, και κατάργηση θανατικής ποινή παγκοσμίω. Αυτά ζητούν οι πολίτες. Να είμαστε συνεπείς και αποτελεσματικοί στην υπεράσπιση αυτών των αξιών και αυτό θα πρέπει να στέλνει ένα σαφές μήνυμα στους πολίτες ότι η φωνή τους γίνεται ακουστή. Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ και πάλι την Αντιπρόεδρο, την κυρία Αντζελίλη, για την πρωτοβουλία αυτή. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι βέβαιο ότι ο συνάδελφός μου Ότμαρ Κάρας θα συμπληρώσει την εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί η επικοινωνία να βοηθήσει την πρόθεση ισότητας των φίλων. Ευχαριστώ πολύ. Ladies and gentlemen, uh, friends. Uh, Κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι, να ευχαριστήσω καταρχήν την Αντιπρόεδρο την κυρία Αντζελίλη και να ευχαριστήσω επίση τον Πρόεδρο Γκούστασον της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ίση Εκπροσώψη για την, για την πρωτοβουλία αυτή. Και μας καταδεικνύουν τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν καλύτερα στα θέματα αυτά. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν για την υποστήριξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και για την προσήλωσή σας στα θέματα αυτά. Θέλω και εγώ να προσυπογράψω αυτό το οποίο λέτε, ότι ένα άμεσα εκλεγμένο θεσμικό όργανο, άμεσα εκλεγμένο από τους πολίτες, όχι μονάχα θα πρέπει να ακούσει την άποψη των πολιτών, αλλά θα πρέπει περαιτέρω και να δρά ακολουθώντας αγνώμονα τις ε, επιθυμίες και τις ανάγκες των πολιτών. Και αυτή είναι και η υποχρέωσή μας όχι μόνο να αναλύουμε και να κάνουμε διαγνώσεις αλλά και να δρούμε ιδίως σε μια εποχή οικονομικής κρίσης και κρίσης εμπιστοσύνης στην πολιτική τάξη. Πρέπει να αναρωτηθεί κανείς αν είναι πιο σημαντικό να συζητάμε για νομικά και οικονομικά ζητήματα ή για αξίες. Κατά την άποψή μου δεν είναι αμοιβαίως αποκλειόμενα αυτά τα δύο. Πιστεύουμε ότι σε μια εποχή κρίσης είναι σωστό και πρέπει να αναστοχαζόμαστε και για τις αξίες γιατί αυτό μας επαναφέρει στην βάση της σκέψης μας και του ευρωπαϊκού εγχειρήματο και ιδίως σε καιρούς κρίσης οι αξίες μας δοκιμάζονται και τίθενται υπό αμφισβήτηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οργανώνει τέσσερις εκστατείες επικοινωνίας που εστιάζουν σε τέσσερις κέρυες αξίες. Την ισότητα των φύλων, την πολιτιστική πολυμορφία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την έννοια της ευρωπαϊκής ηθαγένειας. Και οι τέσσερις αυτές είναι αξίες τις οποίες προωθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να οργανώνει εκδηλώσεις και γεγονότα όπως η σημερινή συνεδρίαση, ώστε να είναι σαφής η ανυποχώρητη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με αυτές τις αξίες όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όταν όμως υπάρχουν προβλήματα με αυτές τις αξίες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί μόνο του να πλησιάσει όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας από τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνθήκη της Λισαβόνας κατέδειξε τη σημασία και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων και την αναβάθμισε. Η συνεργασία μεταξύ του Εθνικού Κοινοβουλίου και των του Ευρωπαϊκού και των Εθνικών Κοινοβουλίων είναι απαραίτητη. Υπάρχουν πολλοί τομεί όπου ακόμα γίνονται προσπάθειες αλληλοεπικαλυπτόμενες και παράλληλες και όχι μέσα στα πλαίσια μιας συνέργειας. Οι εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να συμβάλλουν μαζί με τα γραφεία πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε, στην επίτευξη μιας καλύτερης συνεργασίας. Με τη σημερινή ευκαιρία το, τα γραφεία πληροφορίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορούσαν να είναι και ο χώρος όπου συγκεντρώνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και ανταλλάσσονται με εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων προτού να μεταλαμβαδεύσουν τα τελευταία το μήνυμα προς τους πολίτες. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορούμε να οργανώσουμε μια συζήτηση σε όλα τα γραφεία πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα το οποίο μας απασχολεί εδώ σήμερα και επίσης που συζητήσαμε χθε με ειδικευμένου δημοσιογράφους για να υποστηρίξουμε καλύτερα το έργο μας. Υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν ήδη αναπτυχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να προαχθεί η ισότητα των φύλων και ιδίως σε ό,τι αφορά τις γυναίκες σε θέσεις εξουσίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κατ' επανάληψη υποστηρίξει την θέση του υπέρ των ποσοστώσεων, διότι θεωρεί ότι αυτό θα είναι ένας τρόπος με τον οποίο θα μπορέσει να αυξηθεί ο αριθμός των γυναικών σε διοικητικά συμβούλια που έχουν εποπτικό χαρακτήρα. Ξέρουμε ότι πάνω από 55% όλων των υποψηφίων είναι γυναίκες αλλά αυτό το ποσοστό δεν αντανακλάται στις θέσεις ευθύνης σε διάφορους οργανισμούς για τις γυναίκες. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συνεχίσει να διεκδικεί ένα πιο δίκαιο και καλύτερο τρόπο προώθησης της ισότητας των φύλων και στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο έχουμε ζητήσει την επιβολή ποσοστώσεων σε, με διάφορα νομοθετικά μέτρα η πρόοδος που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής για την ισότητα των φύλων ποικίλει από κάτω μέλος σε κάτω μέλος. Και αυτό διαφάνηκε από τη συζήτηση που έλαβε χώρα προηγουμένω. Αλλά εμείς ως πολιτικοί δεν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ε, εκδίδουμε κανονισμούς και οδηγίες, αλλά θα πρέπει να είμαστε και υπόδειγμα στον τομέα αυτό. Αν εξετάσουμε το δικό μας τομέα, είναι φανερό ότι η πολιτική ακόμα έχει πολύ δρόμο να διατρέξει για τα θέματα αυτά. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας ορισμένα στοιχεία σε σχέση με τις γυναίκες στον πολιτικό στίβο. Είναι αποκαλυπτικά τα στοιχεία αυτά και καταδεικνύουν ότι υπάρχει πολύ περιθώριο βελτίωσης. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως ανέφερε η συνάδελφός μου κυρία Αντζελίδη, 65% των εδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανήκουν σε άνδρες, ενώ 35% μόνο γυναίκες. Σε επίπεδο κρατών μελών είναι ακόμα μεγαλύτερο το χάσμα. 75% των μελών των Εθνικών Κοινοβουλίων είναι άνδρες και μόνο 25% γυναίκες. Δεν υπάρχει ούτε ένα κοινοβούλιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου να υπάρχουν περισσότερες γυναίκες από άνδρες. Θα ήθελα λοιπόν να κλείσω επανεχόμενος σε κάτι που είπε η κυρία Ποδηματά. Κατά μέσον όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι γυναίκες κερδίνουν, κερδίσουν 17,5% λιγότερο από τους άνδρες για έργο ίσης αξίας. Βάσει των στοιχείων του Ευρωβαρομέτρου με την ευκαιρία της ημέρα των γυναικών 8 Μαρτίου του 2012 οι περισσότεροι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή η οποία θα πρέπει να δράσει για να μειωθεί το χάσμα στις αμοιβέ ανδρών και γυναικών. Και θα πρέπει να προωθήσουμε λοιπόν όλο και περισσότερη ισότητα στα δικά μας κοινοβουλευτικά όργανα. Και να πω και κάτι στη μητρική μου γλώσσα, κύριε Πρόεδρε. Εγώ είμαι πρόεδρος μιας κοινωνικής ΜΚΟ, η οποία ασχολείται με κοινωνικά θέματα και θέματα υγειονομικής περίθαλψης. Και γνωρίζω ποιες είναι οι διαφορές στην κοινωνία μας. Στο παρελθόν. Οι γυναίκες είχαν να αντιμετωπίσουν τεράστια μειονεκτήματα στον χώρο εργασίας λόγω των οικογενειακών τους υποχρεώσεων. Σήμερα όμως έχουν αλλάξει οι οικογενειακές συνθήκες, έχει αλλάξει η δημογραφική δομή της κοινωνίας και αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες υφίστανται περισσότερο φόρτο εργασίας διότι έχουν να αντιμετωπίσουν και τη φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων. Είναι οι ίδιες γυναίκες οι οποίες εργάζονται πολλές φορές και οι οποίες είναι πάντα οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις απόρριες της νέας αυτής δημογραφικής εξέλιξης της κοινωνίας μας και των κοινωνικών αλλαγών στον χώρο εργασίας. Ανεξάρτητα οποιαδήποτε νομοθετική ε, ρύθμιση Εάν δεν λάβουμε υπόψη την, ε, τις επιπτώσεις αυτών των νέων προκλήσεων για τις γυναίκες μέσα στα φορολογικά συστήματα και στα συνταξιοδοτικά συστήματα, τότε θέτουμε τις γυναίκες σε μια μόνιμη κατάσταση επιβάρυνσης, η οποία είναι σε βάρος της και η οποία δεν επιτρέπει μια επαρκή ε, ένα, ένα επαρκή βαθμό συμβιβασμού της οικογενειακής και της ε, επαγγελματικής ζωής. Αυτό δεν είναι μονάχα ένα εθνικό καθήκον, είναι συγχρόνως και ένα εγχείρημα που πρέπει να απασχολήσει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο να δημιουργηθεί η απαραίτητη συνειδητοποίηση για το πρόβλημα αυτό και στη μελλοντική στρατηγική να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πείσει τα κράτη-μέλη στο να προχωρήσουν σε αλλαγές στα κοινωνικά συστήματα και συστήματα απασχόλησής τους. Έχουμε πάρα πολλά λοιπόν να πράξουμε. Είναι, δεν είναι λιγότερα, είναι περισσότερα τα καθήκοντά μας και στο μέλλον θα είναι ακόμα περισσότερα και παρά το γεγονός ότι έχουμε προχωρήσει αρκετά, δεν έχουμε φτάσει στο τέλος του δρόμου. Και χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι η Επιτροπή Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ως πρόεδρο ένα άνδρα ο οποίος έχει την σαφή αυτή προσήλωση στα θέματα των γυναικών όπως ο κύριος Γκούσταυσον. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια νομοθετική επανάσταση. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένα όργανα, μέσα, εργαλεία, υπηρεσίες, ευελιξία στην απασχόληση. Χρειάζεται όμως και μια αλλαγή νοοτροπίας. Θα ήθελα μόνο να πω κάτι σε σχέση με τα όσα έλεγε ο συνάδελφος Κάρας. Ότι δηλαδή κάποιες φορές και σχεδόν πάντα τις γυναίκες βαραίνει η οικογένεια. Εγώ προσωπικά σας λέω ότι πολλές φορές που είμαι εδώ στις Βρυξέλλες στο Στρασβούργο που και που και ακόμα και την ώρα που προεδρεύω στις κοινοβουλευτικές εργασίες δηλαδή μπορώ να κάνω απολύτως τίποτα Κάποιος από την οικογένεια μου στέλνει ένα μήνυμα στο κινητό να μου πει υπάρχει το τάδε πρόβλημα. Ε, τι να πω, πρακτικό, οργανωτικό, τι να κάνουμε και εγώ από το τηλέφωνο πρέπει να απαντήσω. Γιατί πολύ συχνά στο σπίτι, άμα δεν είμαι εγώ, δεν λειτουργεί τίποτα και με έχουν ως σημείο αναφοράς για όλα τα πρακτικά ζητήματα. Χρειάζεται λοιπόν και αυτή η αλλαγή νοοτροπίας. Εντάξει, μπορεί να είναι κανεί αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά στα πρακτικά συγκεκριμένα θέματα τη οικογένεια πάντα είναι οι γυναίκε και υπό οποιασδήποτε συνθήκε ασχολούνται οι γυναίκε. Υπάρχουν τώρα άλλες παρεμβάσεις, η κυρία Λετσόφσκα ή κάπως έτσι. Ευχαριστώ πολύ, ε, ε, κυρία Πρόεδρε. Μου αρέσει πάρα πολύ το θέμα του σημερινού σεμιναρίου, διότι η επικοινωνία στο σημερινό κόσμο είναι πραγματικά ε, ένα πολύ αποτελεσματικό μέσο και εργαλείο για να φτάνει κανείς στον πολίτη. Παντού, όχι μόνο στην Ευρώπη, σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ εύκολο να δούμε, κυρίες και κύριοι, πώς η επικοινωνία σε διάφορα επίπεδα ε, βελτιώνεται η επικοινωνία είναι καλύτερη πολλές φορές και από τους βουλευτές προς τους πολίτες όταν πρόκειται για γυναίκες. Από γυναίκα σε γυναίκα, ενώ από άντρα σε άντρα είναι πιο δύσκολη η επικοινωνία. Ε, γυναίκες πολλές φορές βλέπουν με διαφορετικό τρόπο τα πράγματα και τα διοικητικά και τα οργανωτικά και τα καθημερινά και τα περιγράφουν πολύ καλύτερα από τους άνδρες. Και πολλές φορές βλέπουμε ότι οι γυναίκες έχουν ένα ε, ρόλο που τους αναλογεί που είναι να λύνουν προβλήματα. Ε, και ε, όλα αυτά όμως δεν ενδιαφέρουν τα μέσα ενημέρωσης, γιατί δεν πουλάνε, δεν είναι δημοφιλή. Και πολλές φορές όλα αυτά ε, ε, τα προβλήματα τα λύνουν οι γυναίκες, τα διεκπεραιώνουν και τελικά οι άνδρες είναι εκείνοι που δρέπουν τις δάφνες στα μέσα ενημέρωσης και στον τύπο και στο facebook και παντού. Δηλαδή πίσω από τις αποφάσεις και τις δράσεις κρύβονται γυναίκες, τελικά οι άνδρες όμως αποκομίζουν τους επένους. Και όταν γίνεται λόγος ε, για την κοινωνία, για τους πολιτικούς, για τους δημοσιούς υπαλλήλους, είναι τεράστια ε, η ε, σημασία των μέσων ενημέρωσης. και κυρίως τα εμπορικά κανάλια και τα εμπορικά μέσα που ασχολούνται με την καθημερινότητα των πολιτών και την αναφέρουν και την προβάλλουν. Πολλές φορές βλέπουμε λοιπόν ότι για να συνδιαλεγούν με την κοινωνία και να επικοινωνήσουν με την κοινωνία και τα ίδια τα μίντια καλούν άνδρες. Στις τηλεοράσεις μας στην Πολωνία, αλλά πιστεύω και σε άλλες χώρες ισχύει αυτό, υπάρχουν πολλά προγράμματα όπου δεν βλέπεις πουθενά γυναίκα, γιατί δεν καλούν γυναίκες. Γιατί δεν θέλουν να τις ακούνε. Έτσι το ερμηνεύω. Κυριαρχούν οι άνδρες σε αυτά τα προγράμματα και είναι και πολύ μεγάλη η συγκατάβαση και ε, ε, η ε, επικοινωνία μεταξύ τους, αλλά εμείς θέλουμε να βλέπουμε και γυναίκες στη τηλεόραση. Και βέβαια όταν σε κάποια πολιτικά φόρα είναι μόνο άνδρες, αυτό δεν μπορούμε να το αλλάξουμε, αλλά από την κοινωνία μπορούμε να καλούμε γυναίκες άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τα προγράμματα της τηλεόρασης ή άλλα μίντια. Θα πρέπει να υπάρχουν ποσοστώσεις, εκεί συμφωνώ. Όταν γίνεται συζήτηση, ας πούμε ένα debate, να είναι ίδιος αριθμός ανδρών και γυναικών σε ένα πάνελ. μια ποσόστοση, αν δεν είναι 50-50 να είναι 30-40, να φαίνονται οι γυναίκες, γιατί δεν φαίνονται στα μίντια. Και είναι πολύ σημαντικό για τις ποσοστώσεις, ωραία, να γίνονται σεβαστές και μετά τι έγινε, ξεμπερδέψαμε με τις γυναίκες, τους δώσαμε το σωστό τους και τελείωσε. Όχι, θα πρέπει να αξιολογείται ο ρόλος τους, να αξιοποιείται επίσης. Ποτέ δεν θα υπάρξει 100% ισότητα, αλλά τουλάχιστον ακούνε τις γυναίκες. Έστω, ας μην είναι το 50%. Είναι σημαντικό να ακούγονται, να φαίνονται οι γυναίκες και να ε, ανασκουμποθούμε, να αγωνιστούμε για να είμαστε παρούσες και να είμαστε και στο ε, ύψος των περιστάσεων και στο ίδιο επίπεδο με τους άνδρες. Επανειλημμένα οι γυναίκες έχουν αποδείξει ότι όχι μόνο είναι ίσες, είναι και καλύτερες από τους άνδρες αλλά πρέπει να ακούγεται τη φωνή των γυναικών ε, στα δημόσια πράγματα, στο δημόσιο βίο. Και γι' αυτό πιστεύω ότι τα εθνικά κοινοβούλια και τα μέσα ενημέρωσης, όπως είπα προηγουμένως, πρέπει να ε, έχουν αυτό το στοιχείο της ισότητας. Να είναι η πλήρης επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Κάρμεν Κιντανίγια, είμαι η πρόεδρος τη Επιτροπής Ισότητας του, της Βουλής των Αντιπροσώπων στην Ισπανία. Χαίρομαι πάρα πολύ για τη δυνατότητα να είμαι παρούσα ε, μαζί με την ομόλογό μου την πρόοδο της Επιτροπής Ισότητος της Ισπανικής Γερουσίας. Θέλω να σας συγχαρώ λοιπόν για την εκδήλωση αυτή, για το γεγονός ότι έχετε οργανώσει αυτή τη συζήτηση όταν μιλάμε για το θέμα των ποσοστώσεων. Είναι ιδιαίτερα επίκαιρη αυτή η συνεδρίαση. Μιλάμε πάντα για μια πρόκληση που πάντα είναι παρούσα στη ζωή των γυναικών. Είναι πραγματική ισότητα ή παραμένει μονάχα ένα όραμα. Αυτή είναι μια συζήτηση στην οποία πρέπει να εγγύψουμε σήμερα. Μια συζήτηση όπου οι διάφορες κοινοτικές οδηγίες, η τέταρτη διάσκεψη για τις γυναίκες που έλαβε χώρα στο Πεκίνο, όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη μαζί με όλες τις συστάσεις και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το, η ισότητα αντιμετωπίζεται ως, μια, ως ένα δικαίωμα των γυναικών και όχι απλώς ως μια διεκδίκηση. Το ερώτημα λοιπόν να δούμε πού βρισκόμαστε και πού πηγαίνουμε. Έχουμε αντιμετωπίσει τεράστια προβλήματα τα οποία είναι παρόντα στα, στην εργασία, τη, στην θέση, στην ε, ζωή των γυναικών. Πρέπει να μιλήσουμε όμως ακόμα για τη μισθολογική ψαλίδα, για τη βία κατά των γυναικών, για, το λεγόμενο, για τη λεγόμενη κρυστάλλινη οροφή σε σχέση με τη συμμετοχή των γυναικών στην οικονομική και πολιτική ζωή, για το γεγονός ότι οι γυναίκες πλήττονται με ιδιαίτερο τρόπο από την οικονομική κρίση η οποία σοβεί στην ε, παγκόσμια ε, σκηνή και ιδίω σε ορισμένε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι λοιπόν ο ρόλο των γυναικών, ποια αντιμετώπιση θέλουμε να έχουμε σε δύο επίπεδα που συζητάμε. Από τη μια μεριά αντιμετωπίζουμε το θέμα των γυναικών στα μέσα ενημέρωσης. Επίσης, μιλάμε για τις γυναίκες σε επίπεδο ευθύνης, στην πολιτική ζωή, στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων η θέση των γυναικών στις, στα μέσα ενημέρωσης. Μα εκεί οι γυναίκες είναι απούσες. Όταν οι γυναίκες κάνουν μία συνέντευξη τύπου, θα πρέπει αυτή η συνέντευξη τύπου θα πρέπει να έχει κάτι το κοσμοϊστορικό, το εντυπωσιακό, για να μπορέσουν να ασχοληθούν μαζί μας τα μέσα ενημέρωσης. Γι' αυτό είναι απαραίτητο οι κοινοβουλευτικοί, οι βουλευτές και οι γερουσιαστές όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προβαίνουν σε περισσότερες συνεντεύξεις τύπου για μια μεγαλύτερη συνειδητοποίηση των προβλημάτων των γυναικών. Όπως τα κοινοβούλια προωθούν νόμους, θα πρέπει να το παρουσιάζουμε, ότι οι νόμοι αυτοί αλλάζουν την ζωή και την καθημερινότητα των γυναικών. Το κάνουμε αυτό στην Ισπανία. Όλες οι κοινοβουλευτικοί που είναι μέλη της Επιτροπής των Επιτροπών Ισότητος στη Βουλή και στη Γερουσία της Ισπανίας κάνουμε μια ιδιαίτερη προσπάθεια να είμαστε παρούσες στα μέσα ενημέρωσης, να μεταφέρουμε τα στοιχεία της συζήτησης στο Κοινοβούλιο στα μέσα ενημέρωσης, να κάνουμε διασκέψεις τύπου για θέματα άνησης αμοιβή. Όταν μιλάμε για την η ε, οικογενειακή ζωή και την επαγγελματική ζωή και την συμφιλίωσή τους που είναι ένα θέμα ακόμα εκρεμές και για τους άνδρες και τις γυναίκες αυτό είναι κάτι το οποίο το τονίζουμε γιατί οι γυναίκες είναι υποχρεωμένες να επιλέγουν μεταξύ του να είναι μητέρες και του να είναι ενεργές στην πολιτική ζωή όπως πολύ σωστά έλεγε η αντιπρόεδρος η κυρία Αντζελίλη Πολλέ φορές πρέπει να προεδρεύει μια συνεδρίαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενώ ο γιο της έχει ένα οικογενειακό πρόβλημα και ζητάει τη βοήθειά της. Εξακολουθεί λοιπόν να παραμένει η ζωή μας μέσα σε μια πατριαρχική δομή όπου οι γυναίκες δεν συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων και βλέπουμε να έχουμε συνέχεια εμπόδια στο δρόμο μας. <clears throat> Συγχρόνως θα πρέπει να πράξουμε όλα αυτά τα οποία είναι ε, απαραίτητα και δυνατά και συμφωνώ με τον κύριο Γκούσταυσον απόλυτα ότι σε μια τέτοια στιγμή οικονομική κρίση δεν πρέπει να φέρουν το βάρος αυτή της κρίσης οι γυναίκες. Η οικονομική αυτή κρίση θα πρέπει να είναι η ευκαιρία να τονίσουμε περισσότερο την παρουσία των γυναικών στα μέσα ενημέρωση. Γιατί οι γυναίκε έχουν να υποβάλουν και εναλλακτικέ προτάσει <clears throat> για να μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση και πρέπει εμεί να παίξουμε ένα ηγετικό ρόλο σε μια πολύ δύσκολη στιγμή στη ζωή των χωρών μας. Κάτι ακόμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μετά από το γεύμα θα μιλήσουμε για το ρόλο των γυναικών στην πολιτική. Εγώ ενδεχομένως θα πρέπει να φύγω γιατί πρέπει να είμαι στο Συμβούλιο της Ευρώπης αυτό το απόγευμα όπου στις 7 η ώρα θα πρέπει να λάβω μέρος σε μια συζήτηση για την ελευθερία της παιδείας. Θέλω να σας δώσω όμως το εξής στοιχείο. Το 1995 έλαβε χώρα η τέταρτη συνδιάσκεψη για τα θέματα των γυναικών στο Πεκίνο που ήταν ορόσημο για τα θέματα των γυναικών. Το 1995 στον κόσμο οι γυναίκες στα κοινοβούλια σε παγκόσμιο επίπεδο ήταν μόνο 11%. Τώρα το 2012 είμαστε το 18%. Μόνο 7% είναι η διαφορά στα παγκόσμια κοινοβούλια. Αυτή είναι η αύξηση στη συμμετοχή στα κοινοβούλια. Στην Ισπανία βέβαια έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια και οι γυναίκες στην Βουλή και στη Γερουσία είναι το 36% πια. Στην Ισπανική κυβέρνηση οι υπουργοί που είναι γυναίκες είναι το 42%. Στις, ε, στα κοινοβούλια των αυτόνομων περιοχών της Ισπανίας σε ορισμένα κοινοβούλια οι γυναίκες ξεπερνούν, σε ορισμένα αυτόνομα κοινοβούλια ξεπερνούν το 50%. Παρ' όλα αυτά, στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων δεν είναι ακόμα επαρκώς εκπροσωπημένες. Πρέπει να πούμε ότι στην Ισπανία 70% των επιχειρήσεων έχουν μόνο 11% γυναίκες. Να σας δώσω και μερικά ακόμα στοιχεία. 60% των πανεπιστημιακών είναι γυναίκες, ενώ 40% οι άνδρες. 8% στα υψηλότερα διευθυντικά στελέχεια. 5% των προέδρων οργανισμών. Γιατί μιλάμε λοιπόν για ισότητα όταν έχουμε ενώπιόν μας μια κατάσταση ανισότητας. Πρόκειται λοιπόν για το πρόβλημα ότι οι γυναίκες δεν φτάνουν σε επίπεδο λήψης αποφάσεων. Ακριβώς γιατί πρέπει να επιλέξουν μεταξύ της οικογενειακής τους ζωής και της επαγγελματικής τους ζωής. Γιατί εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη ε, και αξιοκρατίας. Έχουμε ένα νόμο ισότητα το 2007, όπου, και αυτό ίσως πρέπει να συζητήσουμε και εδώ, Βάσει του νόμου αυτού τα διοικητικά συμβούλια είναι υποχρεωμένα να εξασφαλίσουν βαθμία την αύξηση του αριθμού των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Θα πρέπει να μιλήσουμε λοιπόν για αυτό το θέμα και να δούμε πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να προσκαλέσει τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς βέβαια υποχρεωτικό χαρακτήρα, αλλά προαιρετικά να δημιουργήσει συστήματα, κίνητρα, μεγαλύτερο ενδιαφέρον των ε, μέσων ενημέρωσης. Στοιχεία λοιπόν τα οποία θα εξασφαλίσουν ότι μπορούν σιγά σιγά οι γυναίκες να σπάσουν αυτό το φράγμα της ανισότητας και να συμμετέχουν όλο και περισσότερο στον επιχειρηματικό κόσμο που είναι τόσο σημαντικός λόγω της κρίσης και όπου περισσότερο από ποτέ χρειαζόμαστε την ηγεσία των γυναικών όχι μονάχα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε όλο τον κόσμο. Σήμερα λοιπόν συζητάμε για μια ανισότητα που εξακολουθεί να υπάρχει μετά από τη συνθήκη της Λισαβόνας, μετά από όλες αυτές τις παγκόσμιες διασκέψεις για τα δικαιώματα των γυναικών έχουμε και πάντα ακόμα ακόμα μια κατάσταση ανισότητας. Κύριε Ούσταυσον, η Ισπανία έχει ένα υφυπουργό ο οποίο είναι αρμόδιος για τα θέματα ισότητας. Γιατί ακριβώς πρέπει να δούμε την πολυπλοκότητα αυτού του θέματος της ισότητας. Την ισότητα αυτή που είναι μια πολύπλοκη και πολύ μορφή ε, διεκδίκηση και γι' αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω για τη βοήθειά σας σε αυτό το δύσκολο δρόμο. Σα ευχαριστώ. Έχουμε ακόμα τέσσερι ομιλητέ. Στην πράξη πρέπει εμεί να φύγουμε από την αίθουσα εντό τεσσάρων λεπτών. Μπορούμε να ζητήσουμε από τους διερμηνείς ευγενικά να μας δώσουν λίγο χρόνο παραπάνω, αλλά θα παρακαλέσω όσους θα πάρουν το λόγο από εδώ και μπρος να ε, είναι σύντομοι, γιατί θα έχουμε και το απόγευμα εξάλλου, όπου θα μπορέσετε και πάλι να πάρετε το λόγο αν θέλετε. Θα δώσω λοιπόν το λόγο πρώτα στον κύριο Σαφ. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ. πολύ. Jean-Paul Σαφ, λέγομαι. Είμαι άνδρας βέβαια, όπως βλέπετε, και θα επιτρέψω στον εαυτό μου να παρέμβω εν συντομία. Έρχομαι από το Λουξεμβούργο και είμαι πρόεδρος εκεί της Επιτροπής του Κοινοβουλίου τη Λουξεμβούργου για την οικογένεια, την νεότητα και την ισότητα ευκαιριών. Τα θέματα αυτά που ενδιαφέρουν τις γυναίκες στην κοινωνία και πιστεύω και εγώ ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει συνειδητοποίηση και κινητοποίηση των γυναικών. Βέβαια, από αυτά που βλέπω σε αυτή την αίθουσα, βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή των γυναικών και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Και θα ήθελα να σταθώ σε κάτι που αναφέρατε κυρία Πρόεδρε για το θέμα του συμβιβασμού της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Θα μπορώ να μιλήσω προσωπικά. Θα ήταν χρήσιμο να υπάρχουν και προγράμματα τα οποία να έχουν σαν ομάδα στόχου όχι τις γυναίκες αλλά τους άνδρες. Ακριβώς για το θέμα αυτό της συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Οι άνδρες δεν είναι άμυροι ευθυνών για το γεγονός ότι οι γυναίκες έχουν ένα υπερβολικό φόρτο καθηκόντων. Για να υπάρξει μια επίτευξη ισότητας θα πρέπει να ενθαρρυνθούν και οι άνδρες ώστε να δώσουν στη γυναίκα τους ή στις γυναίκες γενικά περισσότερο χώρο για να μπορέσουν να πέσουν ρόλο στο δημόσιο στίβο. Αυτό σημαίνει ότι οι άνδρες θα πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερες ευθύνες στον κοινωνικό χώρο και στον χώρο της οικογένειας. Είναι λοιπόν και αυτό, αν θέλετε, ένα θέμα επικοινωνίας και ένα θέμα κοινωνικής ε, ε, συμμετοχή των ανδρών που θα πρέπει και αυτό να μπει στο θεματολόγιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Λούλινγκ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πάρα πολύ σύντομα. Πρέπει να πω ότι αισθάνομαι τουλάχιστον 40 με 50 χρόνια νεότερη. Γιατί τόσα χρόνια αγωνίζομαι για την ισότητα των ευκαιριών ε, ανδρών και γυναικών. Ε, πάντα τους ίδιους θρήνους ακούμε και οδυρμούς όλα αυτά τα χρόνια. Και πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν μερικές ε, διεκδικήσεις που παραβιάζουν ανοιχτές θύρες. Ακούσαμε πάλι για την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ε, και να δείτε νόμους που έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το 1975 για αυτά τα θέματα ισότητας αμοιβών αδρό και γυναικών. Πλήρες οπλοστάσιο και είναι πάρα πολύ καλές αυτές οι οδηγίες οι οποίες όμως θα πρέπει να εφαρμόζονται σε επίπεδο κρατών μελών. Ε, γνωρίζω ότι εδώ η Επιτροπή Γυναικών του Κοινοβουλίου πάντα διεκδικεί μεταρρυθμίσεις, αλλά πρέπει να σας πω ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις έγιναν όταν ήμασταν λιγοστές γυναίκες. Ε, αυτή η νομοθεσία υπάρχει, είναι καλή, αλλά πρέπει να εφαρμόζεται. Και δεν ξέρω, ας πούμε, το, να αμφισβητείς αυτές τις οδηγίες, 27 κράτη-μέλη, μπορείς να καταλήξεις σε μια τόσο καλή νομοθεσία όσο αυτή που έχουμε εγώ το έχω ζήσει. Πρέπει να τη χρησιμοποιούμε, να την υλοποιούμε. Βέβαια, είπαμε τώρα για τη μισθολογική ψαλίδα, πόσο αμείβονται οι άνδρες, πόσοι οι γυναίκες. Όλα αυτά είναι μέση όρη. Μέση όρη δεν λένε τίποτα. Γνωρίζω και άνδρες που κάνουν την ίδια δουλειά με άλλους άνδρες και κερδίζουν λιγότερα. Ένας ε, οδηγός λεωφορείου στη χώρα μου, πούλμαν ιδιωτικού, κερδίζει πολύ λιγότερα από ένα οδηγό λεωφορείου δημοσίου. Λοιπόν, οι γυναίκες μπορεί να υφίστανται διακρίσει στην εταιρεία τους ε, σε σχέση με τους άνδρες, αλλά να τους ζητείτε να πάνε να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Και εμείς το κάναμε αυτό. Και εγώ έχω συνεισφέρει και σε κάποιες από τις δίκες τις οποίες τελικά κερδίσαμε. Εκατοντάδες είναι τα εκατομμύρια ε, τη δεκαετία του 70 και του 80 που πληρώθηκαν και μάλιστα αναδρομικά στις γυναίκες στο Λουξεμβούργο, στις δημοσίες υπαλλήλου, διότι το διακρίσεις, παράδειγμα σε ό,τι αφορά ε, το επίδομα οικογενειάρχη. Εγώ ε, έκανα δικαστήριο με κάποιες ε, γυναίκες ε, που δούλευαν στην τοπική αυτοδιοίκηση και ε, αμείβαν το λιγότερο και κέρδισαν αναδρομικά 25 εκατομμύρια και ήρθαν στο γραφείο μου με σαμπάνιες. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην εργασία, την κοινωνική ασφάλιση, έχουμε νόμους, αλλά θα πρέπει να ζητάτε να εφαρμόζονται εσείς στις χώρες σας. Δεν χρειάζεται μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ούτε θα σας βοηθήσει αυτή εάν και πάλι δεν την αξιοποιείτε και δεν την εκμεταλλεύεστε, γιατί υπάρχει η κοινωτική νομοθεσία και είναι και καλή σε όλους τους τομείς αυτούς και σε ό,τι αφορά τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ε, σταματώ εδώ και ε, μην λέτε ποτέ ότι δεν έχουμε τίποτα και θα πρέπει να εφεύρουμε τα πάντα. Τον τροχό δεν χρειάζεται να τον επαναφεύρουμε στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την Ισότητα Αμοιβών Απλώς χρειάζεται σωστή εφαρμογή και υλοποίηση των νόμων. Ehm, Σας ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλες δύο παρεμβάσει. όμως θα ήθελα να ρωτήσω τόσο την κυρία Τούμο, και την κυρία Μανατίδου ε, αν μπορούν να παρέμβουν αργότερα έτσι ώστε να έχουν και περισσότερο χρόνο για να κάνουν τις παρεμβάσεις τους και να ζητήσω την Αντιπρόεδρο Ποδηματά και τον Αντιπρόεδρο Κάρας αν θέλουν να κάνουν μια τελευταία παρέμβαση ε, καταλήγοντας εδώ, τελειώνοντας και ευχαριστώ και τους διερμηνείς καθώς και την Γενική Διευθύντρια Διερμηνίας την κυρία Κοσμίδου που είναι υπεύθυνη για τη διερμηνία και για τη βοήθεια που μας έδωσε για τη διοργάνωση τούτης εδώ της ε, διάσκεψης. Thank you very much. Grazie, Roberta. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ε, Ρομπέρτα. Δύο λόγια θα πω μόνο στα ελληνικά, στη μητρική μου γλώσσα. Uh, not, uh, In my function as vice. Όχι υπό τη ιδιότητα τη Αντιπροέδρου που με αρμόδια για την επικοινωνία, αλλά ω μέλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ω γυναίκα Ευρωβουλευτή. Ε, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συζήτηση που γίνεται. Ε, θέλω να πω το εξής. Ε, μιλήσαμε για τις ε, πρακτικές που ισχύουν, για την ομοθεσία που ισχύει στο ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη συμμετοχή των γενικών στην πολιτική, ε, την εκπροσώπηση των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όπως σωστά επισημάνθηκε από πολλούς συναδέλφους και πολλές συναδέλφισες, αυτό αντικατοπτρίζει ένα μέσο όρο. Ο μέσος όρος δεν έχει να κάνει με την πραγματικότητα που υπάρχει στα διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πραγματικότητα είναι ότι σε αυτά τα ζητήματα της ισότητας των φύλων υπάρχουν τεράστιες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών. Το 75% κατά μέσο όρο συμμετοχή των γυναικών στα εθνικά κοινοβούλια ε, ανδρών και 25% γυναικών σε ορισμένα κράτη μέλη ε, σημαίνει 50-60% συμμετοχή γυναικών και 40% συμμετοχή ανδρών σε λίγα κράτη μέλη. Σε άλλα κράτη μέλη η αναλογία είναι πολύ δυσμενέστερη από αυτό το 75-25%. Ο συνάδελφός μου, ο αντιπρόεδρος Κάρας, επεσήμανε πολύ σωστά στην παρέμβασή του τις επιπτώσεις της δημογραφικής εξέλιξης στην Ευρώπη στα ζητήματα της ισότητας των φύλων. Συναδέλφοι από την Ελλάδα, την Ισπανία, αλλά και ο ίδιος ο πρόεδρος της Επιτροπής Γυναικών, η αντιπρόεδρος Αντζελίλη, αναφέρθηκαν στις επιπτώσεις της ίδιας της κρίσης στα ζητήματα της ισότητας. Και μία από τις επιπτώσεις αυτές αφορά στον πολύ ορατό κίνδυνο το χάσμα αυτό στο οποίο αναφέρθηκα οι τεράστιες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών στα θέματα της ισότητας να γίνουν ακόμα μεγαλύτερες εξαιτίας της κρίσης ακριβώς διότι ε, η αποδόμηση του, ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου ε, οι δραστικές περικοπές που εφαρμόζονται σε μια σειρά χώρες όχι πια μία και δύο στα ζητήματα της κοινωνικής πολιτικής έχουν ευθεία επίπτωση και αντανάκλαση στις δυνατότητες των γυναικών όχι μόνο στην πολιτική αλλά στην επιχειρηματικότητα στην εργασία είναι όλα αυτά ζητήματα άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. εγώ εκείνο που θα ήθελα λοιπόν να πω όχι ως συμπέρασμα ως παρότρινση περισσότερο είναι το εξής ε, ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε σήμερα στην Ευρώπη προκειμένου να βγούμε από αυτή την κρίση είναι οι κατακαιρματισμένες και εθνοκεντρικές λογικές. Πιστεύω ότι ε, ως γυναίκες αλλά και ως άνδρες που δεσμεύονται και σέβονται τις αξίες και τις αρχές της ισότητας όπως είναι πολλοί συναδελφοί μας σήμερα μέσα σε αυτή την αίθουσα αλλά και έξω από αυτή θα πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα και μπορούμε να το κάνουμε αυτό της δικτύωσης μεταξύ μας στο ευρωπαϊκό επίπεδο της συνεννόησης μεταξύ μας στο ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε αυτά που ισχύουν ως δυνατότητες σε επίπεδο κοινοτικής νομοθεσίας όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Λούλινγκ πριν να μπορέσουν να δημιουργήσουν στην πράξη μια ευρωπαϊκή κουλτούρα στα ζητήματα της ισότητας που να ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη και ε, να γίνεται όπως το κάνουμε με μια σειρά άλλες πολιτικές στα ζητήματα για παράδειγμα της κοινή αγροτικής πολιτικής όπως ξέρετε ε, εφαρμόζουμε τον έλεγχο υγείας το health check μπορούμε να το κάνουμε αυτό και για τα ζητήματα της ισότητας εάν μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες της και τις προϋποθέσεις για έναν τέτοιο ευρωπαϊκό συντονισμό και για έλεγχο και επανέλεγχο σε σχέση με τα βήματα που γίνονται στο εθνικό επίπεδο νομίζω ότι θα έχουμε κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την ε, σωστή κατεύθυνση. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ε, βέβαια εδώ κανονικά δεν θα έπρεπε να έχει το τελευταίο λόγο ένας άνδρας σε αυτή τη διοργάνωση, <laughs> αλλά επιτρέψτε μου να πω μερικά λόγια ε, διευκρινιστικά. Το τηλέφωνο του παιδιού στο Προεδρείο ε, μπορεί να χτυπήσει και να είναι και άνδρας ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων, δεν χρειάζεται να είναι η μαμά του. Είναι πολύ σημαντικό να φτιάξουμε μια κοινωνία ε, που τα παιδιά να μπορούν να τηλεφωνούν και στους δύο γονείς ανεξάρτητα με το που βρίσκονται εκείνη τη στιγμή ο καθένας. Και δεν επιτρέπεται ε, ένα τηλέφωνο που χτυπάει ενός παιδιού να θεωρείται ενόχληση ή προσβολή, αλλά είναι ανάγκη να απαντήσεις. το θέμα δεν είναι η οδηγία, η κανονισμός. Αυτό δεν λύνεται με κανόνες. Είναι τι αξίες έχει το παιδί και πώς συμπεριφερόμαστε στην κοινωνία μας. Και πώς αντιμετωπίζουμε ένα τέτοιο τηλεφώνημα. Θεωρείται ζημιά, ε, ε θεωρείται καλό, το δεχόμαστε. Ένα δεύτερο που ακούστηκε. Συχνά ε, γίνονται συζητήσεις στα μέσα ενημέρωσης και συμμετέχουν μόνο άντρες. Από τη χώρα μου μπορώ να σας πω ότι το σημαντικότερο κατά κανόνα στα μέσα ενημέρωσης είναι υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ των κομμάτων και όχι μεταξύ των φίλων. Και το ερώτημα είναι τι ρόλο παίζουν τα πολιτικά κόμματα στα μίντια. Πρόκειται για τα περιεχόμενα ή για το κομματικό συμφέρον τι εικόνα δίνει μια συζήτηση ή ποια είναι η ουσία της συζήτησης. Και απέναντι στο ε, κομματικό ε, θέμα και τοποθέτηση. Και ε, το θέμα αυτό δεν είναι μόνο για τα μίντια, αλλά ποιον ορίζουν τα κόμματα, ποιος εκπροσωπεί τα κόμματα στη δημόσια συζήτηση, ποιος εκπροσωπεί τα θεσμικά όργανα και τους θεσμούς γενικότερα στη δημόσια συζήτηση. Και είναι πιθανό εμείς ως κόμματα συχνά να επεμβαίνουμε και απέναντι σε θέματα ισορροπίας φίλου λόγω ε, ενός κομματικού συμφέροντος που θα έχουμε από τα μέσα. Παρά τα μέσα ε, θα πρέπει εκεί να δούμε ποιος εκπροσωπεί σε ποιο φόρουμ. Γιατί υπάρχει συχνά μια σχέση μεταξύ της δημόσιας εικόνας στα μίντια και της ε, αξίας ε, και τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τα κόμματα τα ίδια, ποιον στέλνουν. Στη συνέχεια, απαγορεύονται οι διακρίσεις. Αυτό είναι βασική αρχή και αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτή η αξία μας θα πρέπει να επιβάλλεται και να χρησιμοποιείται ως μέσο και ως εργαλείο για να διαλύονται οι φυστάμενες διακρίσεις. Αν δεν αλλάξει όμως η δημόσια συνειδητοποίηση, αν δεν αλλάξει ο τρόπος ενημέρωσης και ο τρόπος επικοινωνίας για τις διαφορές που υπάρχουν και για τα αίτια των διαφορών αυτών, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε ένα τον άλλον, δεν πρόκειται να αποφύγουμε ε, τη νομοθεσία, αλλά δεν πρόκειται να έρθει και η κατανόηση γιατί χρειάζονται νόμοι. Το θέμα δεν είναι ποσοστιαίο, πόσοι ε, άνδρες και πόσες γυναίκες. Εντάξει, αυτό το φροντίζουμε, αλλά θα πρέπει να κάνουμε και πρόοδο εδώ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ένα θέμα επικοινωνία. Και να, να πούμε ποια είναι τα αίτια που οδηγούν σε αυτές τις διακρίσεις και εκεί θα πρέπει να αρχίσουμε για να αλλάζουμε την εικόνα στην κοινωνία τον τρόπο αντίληψης έτσι ώστε τα μέσα και τα μέτρα που θέλουμε να επιβάλλουν να μπορούν να επιβληθούν καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ για την αφοσίωσή σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σίγουρα αναλαμβάνει εδώ την ε, αρμοδιότητα να ε, διαλύσει τις ε, διακρίσεις και να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία. Ευχαριστώ και καλή σας όρεξη. Σας ευχαριστώ κύριε Ποδηματάκη, κύριε Κάρας και για τη μελλοντική σας ε, δέσμευση για ενημέρωση για τα δικαιώματα των γυναικών, για την επίτευξη της ισότητας των φύλων. Θα τα πούμε εδώ στις 2 και 4. Ε, έχουμε ένα σύντομο γεύμα στο ε, σαλόνι υπαριθμών 4.